Euh, Colleagues, I apologize for the delay. Συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι για την καθυστέρηση. Είμαστε τα θύματα της απεργίας και καταλαβαίνετε όλοι γιατί είναι πιο ισχνή η παρουσία στη σημερινή συνεδρίαση. Μόλον τούτο θα πρέπει να ξεκινήσουμε το έργο μας. Πρώτα με την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν έχετε αντίρρηση μπορούμε να ότι έχει εγκριθεί η ημερησία διάταξη. Ευχαριστώ. Και έχω τώρα κάποιες ε, ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι θα κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση αύριο το πρωί για να συνεχίσουμε τις ακροάσεις με τους προτινόμενους υποψηφίους για τη θέση του επικεφαλής του ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης Σήμερα θα ακούσουμε τον υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου και οι άλλοι υποψήφοι θα ακροαστούν αύριο το πρωί. Θα έχουμε και μια έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα σημεία. Έκθεση για τα φορολογικά ετήσια ψηφοφορίες για τους ε, υποψηφίους για τις διάφορες θέσεις στο ενιαίο Ταμείο Εξυγένσης, ψήφιση για την αίτηση αντίρρησης και επίσης η πρόταση για μη κατάθεση ε, εξαίρεσης ή αντίρρησης για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και την Οδηγία για την ε, Ανάκτηση και την Εξυγίανση. Και ο κύριος Πάντοαν, ο πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, θα ε, είναι παρόν. Έχουμε λοιπόν επίσης και νέα στοιχεία για τους τριγωνικούς διαλόγους. Πρώτα τα καλά νέα. Έχουμε καταλήξει σε πολιτική συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Στατιστικό Τρίλογο με την βοήθεια της Ιταλικής Προεδρίας του Αρμόδιου Επίτροπου για τα θέματα της Eurostat και επίσης με την υποστήριξη του κ. Μπαγέτο και των ισχυωδών συγητών είμαστε πια σε θέση να ψηφίσουμε μια, μια πρώιμη συμφωνία δεύτερης ακρόασης για ένα σημαντικό θέμα το οποίο χάρη και στην προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξασφάλισε ότι η επικεφαλής της Eurostat θα εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής μας αμέσως μετά την, ε, τον διορισμό του ή της, ώστε να μας παρουσιάσει τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών <clears throat> και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η η δυνατότητα της ε, έρευνας στα εθνικά στατιστικά συστήματα για να μπορεί να αποφευθεί η απάτη σε ό,τι αφορά την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τελικά είναι νομίζω θετικό το αποτέλεσμα του τριγωνικού διάλογου. δεύτερος τριγωνικός διάλογος, πολυμερείς ανταλλαγές. Είχαμε μία συζήτηση που έλαβε χώρα στι 4 Δεκεμβρίου. Δυστυχώ οι θέσει των θεσμικών οργάνων αποκλίνουν ακόμα, είναι ακόμα από μεμακρυσμένε. Στείλαμε ένα σαφές μήνυμα ζητώντα από το Συμβούλιο να κάνει την απαραίτητη κίνηση σε πολιτικό επίπεδο που θα μας επιτρέψει να κλείσουμε με θετικό τρόπο αυτό το σημαντικό τριγωνικό διάλογο. ω γνωρίζετε, ο κύριος Θάλμπα είναι ο εισηγητής. Και τέλος έχω κάτι να πω σε σχέση με τη διαδικασία για την αντιμετώπιση του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν το 2015. Πρέπει να συζητήσουμε με την Κομισιόν στα πλαίσια της Συμφωνίας Πλαισίου. Περιμένουμε να υπάρξει μια απόφαση και ως Κοινοβούλιο θα δώσουμε και εμείς την άποψή μας σχετικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Επιτρόπου του κ. Χίλ και του Αντιπρόεδρου κ. Τιν Μέρμανς και λάβοντας υπόψη και τη σημασία που είχε τον αντίκτυπο που είχε το θέμα αυτό στα μέσα ενημέρωση, να υπενθυμίσω ότι η θέση τη Επιτροπή μα που έχει εγκριθεί ήδη από του συντονιστέ, εμεί αναμένουμε από την Κομισιόν να συνεχίσει το έργο τη σε σχέση με όλα τα θέματα, όλου του φακέλου που παραμένουν ακόμα εκκρεμείς και να αποφύγει τον κίνδυνο πρόωρων ανακοινώσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αρνητικά κίνητρα για τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την επίτευξη συμφωνίας. Αυτή λοιπόν είναι θέση της Επιτροπής ΕΚΟ να συνεχίσουμε το έργο για όλα τα θέματα που έχουν παραμείνει εκκρεμή και η αυτοσυγκράτηση σε σχέση με ανακοινώσεις και εμείς επίσης θα δώσουμε μια απάντηση στην ανακοίνωση που προβλέπεται να δώσει η Κομισιόν στις 16 Δεκεμβρίου. Αυτά ως ανακοινώσει του Προέδρου και το μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης που είναι η πρόταση οδηγίας στην έκθεση για την ε, εταιρική διακυβέρνηση και τα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης και την ενεργό συμμετοχή των μετόχων. Είμαστε και εδώ υπεύθυνοι αρμόδιοι για πολύ συγκεκριμένους λόγους ζητήσαμε την εφαρμογή του άρθρου 54 ιδιαίτερα το 2D, 3D, 9α κτλ. Γιατί πρόκειται για θέματα που εμπίπτουν των αρμοδιοτήτων μας. Θα δώσω το λόγο λοιπόν αμέσως στον εισηγητή, τον κύριο Λούτβικσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να αναφέρω ότι τα δικαιώματα των μετόχων και οι υποχρεώσεις τους δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Η συζήτηση σήμερα ε, χαρακτηρίστηκε από μεγάλη πόλωση. Κάποιοι θεωρούν την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταπληκτική και άλλοι ε, άθλια. Πρέπει πάντως να είμαστε πολύ προσεκτικοί πρέπει να εντοπίσουμε τα καλά σημεία της πρότασης και τα λιγότερο καλά. Και θα πρέπει να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά όλα τα επιχειρήματα, να τα διατρέξουμε, να τα αναλύσουμε, ώστε η γνωμοδότησή μας ε, να είναι αιτιολογημένη και να είναι και ενδεδειγμένη φυσικά. Θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ των δύο άκρων αυτών Θέλουμε να έχουμε μια ανοιχτή ευέλικτη συζήτηση στις επόμενες εβδομάδες από κοινού. Νομίζω θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύση και να λύσουμε και τα διλήμματα που προκύπτουν από αυτή την πρόταση. Πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες μας, να έχουμε μία γνωμοδότηση η οποία θα χαρακτηρίζεται από σύγκληση απόψεων γιατί έγινε αυτή η πρόταση. Συμμερίζομαι την ανάλυση των προβλημάτων από πλευρά τη Κομισιόν. Η διοκτησία πολλέ φορέ, οι ιδιοκτήτε δηλαδή τη εταιρείε είναι πολύ παθητικοί τι περισσότερε φορέ. Αν δείτε αυτού οι οποίοι κατευθύνουν, που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, παραδείγματο χάρη, μπορούν να ε, κατευθύνουν με τις αποφάσεις τους, αλλά μπορούν να ωφελήσουν μόνο ορισμένα σκέλη της εταιρείας, όχι συνολικά την επιχείρηση. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πολλές επιχειρήσεις δρούν ε, πάρα πολύ βραχυπρόθεσμα, υπό την έννοια ότι θέλουν να εργάζονται σε τερμηνέα βάση και να έχουν μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων. Άρα η πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση προοπτική χάνεται και μεταξύ άλλων αυτό έχει το αποτέλεσμα να είναι πολύ χαμηλά τα επίπεδα των επενδύσεων. Επίσης, σημαντικά στήματα που πρέπει να επιληθούν δεν επιλύονται και ε, κάποιες φορές δεν λαμβάνονται και οι σωστές αποφάσεις. Αν κάποιος τα βλέπει τα πράγματα ε, με κοντόφερο τρόπο ή πολύ βραχυπρόθεσμα, ε, εστιάζει μόνο στις αποδοχές. Επίσης αυτή η αδράνεια, η βραχυπρόθεσμη προοπτική είναι ένα θέμα. Το 44% των ιδιοκτητών στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο στην Ευρώπη είναι αλλοδαπές και πολλές φορές είναι δύσκολο να είναι κανείς ε, δραστήριος ε, και, να, και διορατικός όταν ε, μιλάμε για διασυνορικές συναλλαγές. Είναι λογικό λοιπόν κατά την άποψή μου να θεσπιστούν στην Ευρώπη κατώτατοι κανόνες για να λειτουργεί καλύτερα στο πεδίο αυτό η ενιαία αγορά. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να βράσουμε με ομαλό τρόπο από τη μια χώρα στην άλλη και αυτός είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για αυτή την κεφαλαία αγορά την ευρωπαϊκή που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα της αδράνης παθητικότητας ή την έλλειψη ενεργών, ενεργής, ενεργούς προσέγγισης και προσήλωσης είναι να δούμε άλλες πτυχές του θέματος, όπως για παράδειγμα τι επενδύσεις γίνονται από συνταξιδοτικά ταμεία π.χ. και άλλους φορείς. Πολλές εταιρείες θα συνεχίσουν την πολιτική τους εκτός αν εμείς αλλάξουμε τα πράγματα. Αν οι διεθνείς επενδυτές και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων δραστηριοποιηθούν περισσότερο και εξετάσουν τα πράγματα πιο μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ θετικέ συνέπειες και για την ίδια την επιχείρηση. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι όσο πιο ενεργοί ε, και προσιλωμένοι είναι οι ε, επενδυτές και οι Διαχειριστέ ε, περιουσικών στοιχείων, ναι δεν θα είναι πανάκι όλων των ζητημάτων, αλλά σίγουρα ε, θα βοηθήσουν τα πράγματα. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, λίγο ευρύτερα την κατάσταση και να δούμε τι μπορούν να συνεισφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φόρε και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για παράδειγμα, οι ομάδες πιέσεων ενό καταναλωτών, το τοπικό περιβάλλοντο στο οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση βέβαια, οι μέτοχοι και οι θεσμικοί επενδυτές είναι ένα σημαντικό κομμάτι όλης αυτής της ε, εξίσωσης. Όχι όμως το μόνο και γι' αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση όλα αυτά έχει κάνει καλή δουλειά σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες. Όμως ε, εκεί που έχω πιο πολλά ερωτηματικά είναι οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. Είναι μια αρχή που ναι, μπορώ να την υποστηρίξω, όμως στο σχέδιο γνωμοδότησής μου θα ασχοληθώ με κάποιες λεπτομέρειες. Δεν πρόκειται να προτείνω ριζικές αλλαγές σε αυτή την πρόταση. Στο σχέδιο γνωμοδότησής μου λοιπόν θα αναφέρω συνοπτικά πέντε πράγματα. Πρώτον, ποιε είναι οι δυνατότητε των εταιριών να αναγνωρίζουν του μετόχου του. Ε. θα ήθελα να έχω μια προσθήκη για να προωθήσουμε το διάλογο μεταξύ μετόχων. Οι εταιρείε οι οποίε έχουν τη δυνατότητα αναγνώριση, ταυτοποίηση των μετόχων θα πρέπει να μπορούν να ενημερώνουν για αυτά τα στοιχεία άλλες εταιρείες, εφόσον ζητηθεί βέβαια κάτι τέτοιο και αυτό θα βοηθά και την επικοινωνία μεταξύ των μετόχων, για να συζητούν τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία. στο μεταλλαγή των στοιχείων με άλλους μετόχους. Έτσι θα έχουμε καλύτερο διάλογο και καλύτερη διακυβέρνηση. Αν δούμε τώρα τους ε, θεσμικούς επενδυτές και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τη δική τους δουλειά, εδώ θα ήθελα μεγαλύτερο άνοιγμα σε σχέση με αυτό που βλέπουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να προωθήσουμε τη διαφάνεια, να υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιεύσουν, να καταρτίζουν ε, πολιτικές για, τις, ε, για τους ιδιοκτήτες, για τις δομές τις ιδιοκτησιακές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια δομή, η οποία όμως είναι κενή με ε. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να προωθήσουμε και την υποβολή αναφορών. Να δούμε τι ε, διάταξη, τι μορφή και σύνθεση έχουν τα χαρτοφυλάκια αυτών των θεσμικών επενδυτών στις ψηφοφορίες, δικαιώματα ψήφου. Και αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει όσοι καθοδηγούν, δίνουν καθοδήγηση για την ψήφο ε, θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε τα σχετικά. Σε ό,τι αφορά τι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίζω ότι οι προτάσει θα πρέπει... Θα πρέπει λίγο τα πράγματα να μπουν σε μία τάξη. Τα περιθώρια που έχουν οι επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από την πολιτική αμοιβών την οποία έχουν ακολουθήσει θα πρέπει να ελέγχεται κάπως καλύτερα και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η άνθρωπο των μετόχων. Πρέπει να υπάρχει ένα δίκαιο περιβάλλον και να γίνει αποδεκτό ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στις αμοιβέ των διευθυντών, γενικών διευθυντών και να δημοσιεύονται φυσικά. Υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την πολιτική αυτή των αποδοχών. Θα πρέπει ίσως να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια όπως είπα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως επίσης και η λεγόμενη κατεπίγουσα πέληση, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα αν τυχόν εμφανιστεί ένα έκτακτο πρόβλημα να διορθωθεί πάρα αυτά. Έχει σημασία αυτό και σε εθνικό όμως να ισχύσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω προτείνει λοιπόν κάποιες ε, ρυθμίσεις να δώσουμε στα κράτη-μέλη σαν παράδειγμα την δυνατότητα να αποφασίζουν αν οι συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών ε, μπορούν να τίθενται και προς έλεγχο από πλευράς των μετόχων πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, εφόσον δηλαδή οι συναλλαγές αυτές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 5% των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε διαφανείς, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και ελπίζω να συμφωνήσουν και οι άλλοι μαζί μου. Στόχος μου είναι να βρεθούν κάποιες κοινέ λύσεις με μεγάλες πλειοψηφίες που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή μας να επηρεάσει τα μάλα. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Ο κύριος Ανδρέας Σουάμπ είναι ω κυριώδης εισηγητής μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα το απόγευμα και μου ζήτησε να παρουσιάσω ορισμένε παρατηρήσει σε σχέση με την έκθεση από τη δική του οπτική γωνία. Θα το πράξω, αλλά φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τον Όλε ιδιαίτερα για το έργο του εξ του Άνδρες Σφάμπ. Κάποιες γενικές καταρχήν παρατηρήσεις ο στόχος της Κομισιόν να εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία των επενδυτών και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς και από το ΕΛ και τον κύριο Σφάμπ αυτό υποστηρίζεται ο στόχος. Πιστεύει ο κύριος Σφάμπ ότι πρέπει να ελεγχθούν ορισμένες πρόνοιες που έχει θεσπίσει η Κομισιόν. Δεν είναι σίγουρος ότι είναι απαραίτητες όλες αυτές οι πρόνοιες, οι ρήτρες που θέτει η Κομισιόν. Υπάρχει στο δίκαιο των ε, επιχειρήσεων μια παράδοση ε, και μια ποικιλία στα εθνικά δίκαια για τις επιχειρήσεις η οποία δεν λαμβάνεται πλήρως υπόψη στην πρόταση της Κομισιόν και ορισμένα στοιχεία αυτής της πρότασης μπορούν να καλυφθούν ήδη από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, για δύο-τρία σημεία κάτι πιο συγκεκριμένα θέλω να πω στο σημείο α, 9α, το δικαίωμα απόφασης για την πολιτική ε, τον των πόνους που δίνονται στα στελέχη. Εδώ θεωρεί ο κ. Σουάμπ ότι η πρόταση της Κομισιόν έχει ένα πάρα πολύ πολύπλοκο πλαίσιο το οποίο δημιουργεί για το θέμα αυτό. Δεν είναι σίγουρος ότι είναι απαραίτητα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση και θα ήθελα να υπάρξει μια προσεκτική εξέταση του αν όλες αυτές οι διατάξεις του άρθρου 9.3 είναι απαραίτητες και αν με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά βελτιώνεται ο έλεγχος των μετόχων πάνω στην επιχείρηση. Ένα δεύτερο στοιχείο, το άρθρο 9β, η απόφαση σε σχέση με την έκθεση που έχει να κάνει με τα, με μπόνους. και εκεί δεν είναι πεπισμένος ο εισηγητής μας ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια απόφαση για το θέμα αυτό, γιατί αυτό ουσιαστικά επαναλαμβάνει την έγκριση που έχει δοθεί προηγουμένως από τους ε, μετόχους, από το Συμβούλιο των Μετόχων. Και επομένως δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνεται αυτό και να υπάρχει δεύτερος έλεγχος και διπλή ρύθμιση της πολιτικής για τα πριμ και τα μπόνους των στελεχών. Αυτό απλώς ε, προκαλεί ένα πρόσθετο κόστος διαχείρισης το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί. Επίσης ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να αναφέρω είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια διακριτική για τις δομές τις οποίες θέλουν να θεσπίσουν σε εθνικό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Τέλος, το σημείο 9 σε. Οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη και η έγκριση που χρειάζεται για αυτές τις συναλλαγές. Εδώ έχει τονίσει ο κύριος Φαμπ ότι πρέπει να υπάρξει η έγκριση των μετόχων, όπως λέει και η πρόταση της Κομισιόν. Αλλά ο τομέας ε, εφαρμογής αυτής της ε, ανάγκης έγκρισης του φαίνεται ότι είναι υπερβολικά ευρύς. Κατά την άποψή του αυτό θα κάνει πιο δύσκολο το έργο των επιχειρήσεων και θα επιβραδύνει την λήψη των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν, επομένως θα έχει τελικά αρνητικό αντίκτυπο στην φυσιολογική λειτουργία των επιχειρήσεων. Τέλος, το σύστημα αυτό δεν θα πρέπει να έχει φυσικά αρνητικό αντίκτυπο στις ε, επιχειρήσεις σε καθημερινό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα να εστιάζεται περισσότερο μονάχα σε συγκεκριμένες συναλλαγές οι οποίες επέχουν ένα κίνδυνο για την επιχείρηση και όχι στο σύνολο των συναλλαγών. Αυτά λοιπόν θα ήθελε ο κύριος Σουάπ να μεταφέρω εξ ονόματός του και αυτό προσπάθησα να πράξω. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος για την ομάδα των συντηρητικών ο κύριος Τέρχο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τον κύριο Φόξ που είναι ο σκιώδης εισηγητής και είναι απόν σήμερα. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την πρόταση του. Αναγνωρίζουμε τα θετικά στοιχεία για την μακροπρόθεσμη συμμετοχή των μετόχων και καλωσορίζουμε πρωτοβουλίες οι οποίες διευκολύνουν τις δραστηριότητες των μετόχων και αυξάνουν τη διαφάνεια. Ο κύριος Φόξ λοιπόν εν πωλής υποστηρίζει τους στόχους της συγκεκριμένης οδηγίας και συμφωνεί ότι η εμπλοκή των μετόχων στην, ε, στην διακυβέρνηση των εταιριών παίζει μεγάλο ρόλο. Συνειδητοποιούμε επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μετόχων και προτύπων μετόχων και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια συνολική σφαιρική αντιμετώπιση κάτω από όποιες συνθήκες διαφορετικές μάλιστα. Η πρόταση αυτή είναι μια πρόταση οδηγίας εναρμόνισης κατελάχιστον ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι αυτά ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν και τις πρακτικές που ακολουθούνται να αποφασίσουν αν η απέτηση ενημέρωσης των μετόχων είναι αναλογική άνω του 5% σε σχέση με τις ε, συναλλαγές. Θεωρεί ο κύριος Φόξ ότι είναι ίσως απαραίτητο να υπάρξουν και κάποιες αποκλήσεις από τον κανόνα έτσι ώστε το καθεστώς να είναι λειτουργικό πέραν των εξαιρέσεων για συναλλαγές από επιχειρήσεις που ανήκουν ε, ολικά σε μια μεγαλύτερη εταιρεία και κάποιες άλλες εξαιρέσεις. Υποστηρίζει ο κύριος Φόξ τις τροπολογίες του εισηγητή για να προστατευτεί η εσωτερική αγορά αντιμετωπίζοντας και τις επιβολές τελών που λειτουργούν στρεβλωτικά για τον ανταγωνισμό σε διαμεθοριακό επίπεδο. Η διαφάνεια είναι σημαντική, αλλά αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θίγει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των νομικών προσώπων και της ασφάλειας των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και θα συμφωνήσουμε με τις επεξηγήσεις του εισηγητή. Η τροπολογία υπάρχει 12 ζητά να υπάρξει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στις δημοσιεύσεις και στην προστασία στοιχείων και στην προστασία των εταιρικών δεδομένων. Ο κύριος Φόξ δεν συμφωνεί απολύτως όμως με τις τροπολογίες 22 και 23. Δεν είναι ιδιαίτερα εξισορροπημένες. Αν και στόχος είναι να καταστήσει τους μετόχους καλύτερα ενήμερους, ε, η καταλληλότητα των ενημερώσεων αυτών, των στοιχείων των ενημερωτικών πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης συνολικά και την πολιτική αμοιβών την οποία ακολουθεί η επιχείρηση ε, και όχι να υπάρχει μια γενική έκθεση για τα πεπραγμένα της επιχείρησης, κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί και λιγότερο χρήσιμο. Θα ήταν λάθος να υποτιμήσουμε ε, ή να αγνοήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχει αυτός ο τομέας. Ε, διαφωνούμε με τις τροπολογίες 4 και 32 όπου αναιρείται το έλεγμα συμμορφώσου ή εξηγήσου. Ε, νομίζω ότι επίσης υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με την πολιτική των αμοιβών ε, και για τις ρυθμίσεις στις οποίες, στα πλαίσια των οποίων οι μέτοχοι, έχουν αποδεχθεί ε, στα ύψη των αμοιβών, τα επίπεδα των αμοιβών. Θα πρέπει λοιπόν η διαφάνεια η οποία εδώ επιζητείται να διευκρινίζει την πολιτική αμοιβών, να είναι κατανοητή η πολιτική αμοιβών της επιχείρησης και να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στις αμοιβέ και τους στρατηγικούς στόχους και επιδόσεις της επιχείρησης. Αυτό ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2013. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Ε, I ευχαριστώ. Δεν βλέπω εδώ εκπρόσωπο των φιλελευθέρων και γι' αυτό θα περάσω στην ΚΟΕ. Ο κύριος Γιέγκας έχει το λόγο. Αυτή η έκθεση αντιμετωπίζει μια σημαντική προβληματική, η οποία είναι ιδιαίτερα εκτενής βέβαια προβληματική και γύρει πάρα πολλά θέματα οικονομικού χαρακτήρα αλλά και ιδεολογικού χαρακτήρα. και φυσικά έχει να κάνει και με το υπόδειγμα χρηματοδότηση που ακολουθείτε και με την εμπιστοσύνη που δημιουργείται στους μετόχους. Επομένω θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα υπόδειγμα το οποίο βασίζεται, το οποίο εστιάζει στους μετόχους και ένα μοντέλο το οποίο εστιάζεται στον συνολικό κοινωνικό αντίκτυπο μιας επιχείρησης. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η έκθεση αυτή ξεκινάει από λανθασμένη εκκίνηση τίθεται το θέμα principal agent, δηλαδή του εντολοδόχου και του εκτελεστή των εντολών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, στο μοντέλο το οποίο βασίζεται στους μετόχους, ουσιαστικά υπάρχει η περίπτωση του εκτελεστή των εντολών, ο οποίος προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την ε, αξία την οποία προσπορίζονται οι μέτοχοι αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι υποχρεωμένος να υιοθετήσει μια μειοαντιμετώπιση αντιμετώπιση σε σχέση με τους μακροχρόνιους στόχους της επιχείρησης και επομένως ακολουθεί μια κοντόφθαλμη λογική. Και αυτό, αυτό θα μπορούσε κανείς να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Θα ήταν ίσως προς το συμφέρον μιας επιχείρησης να επιζητεί το αντίθετο, να επιζητεί να ε, το κέρδος σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και όχι μονάχα σε πρόθεσμο όπως γίνεται. Εν πάση περιπτώσει είναι τρία σημεία τα οποία εδώ θα ήθελα να εξάρω. Το πρώτο στοιχείο είναι ακριβώς η έννοια της στρατηγικής κατεύθυνσης. Με ποιο τρόπο εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε <clears throat> τους μηχανισμούς οι οποίοι παρέχουν κίνητρα τα οποία θα διορθώσουν τη μειοπική κοντόφθαλμη αντιμετώπιση και να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις και οι μετοχή τους θα έχουν μια πιο μακρόπνοη αντιμετώπιση σε σχέση με τις εργασίες των επιχειρήσεων και δεν τους ενδιαφέρει μονάχα το εύκολο, το γρήγορο κέρδος. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κάνει η έκθεση για τα θέματα αυτά. Δεν βλέπω τα, κατά πόσο τα μέτρα τα οποία προτείνονται ε, στην έκθεση θα αλλάξουν αυτή τη βασική κατεύθυνση που είναι κοντόφθαλμη. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσει να υπάρξει κάποια αλλαγή θα πρέπει να υπάρξει ένα πιο κοινωνικό μοντέλο, να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων. Να κατανοήσουμε όλοι ότι η επιχείρηση λειτουργεί σε ένα κοινωνικό χώρο, ότι δρά στον κοινωνικό περίγυρο, έχει επίπτωση στην προσωπική ζωή και τη μοίρα των εργαζομένων, των προμηθευτών, του, της περιοχής όπου βρίσκεται, όλης της κοινωνίας. Γι' αυτό εμείς θα θέλαμε να υπάρξει μια εμβάθυνση της δημοκρατίας, να μην σταματάει η δημοκρατία στις πόρτες των επιχειρήσεων, να υπάρξουν μηχανισμοί οι οποίοι θα εμπλέκουν τους εργαζόμενους στις σημαντικές αποφάσεις της επιχείρησης και να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής κοινότητος, να υπάρχουν χώροι συζήτησης και να υπάρξει μια διευρυμένη συζήτηση, να επιζητείται λοιπόν μια συνένεση σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί η επιχείρηση, επομένως με τον τρόπο αυτό να εμπλέκεται και η επιχείρηση στην κατεύθυνση μιας πιο μακροχρόνιας, μιας πιο ε, μακροπρόθεσμης ε, ανάπτυξης. Τα θέματα τώρα των αμοιβών των στελεχών. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν και κάποια όρια στην ατομική ελευθερία ή την ελευθερία των επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανισότητα κατάφορη μέσα της επιχειρήσεις σε σχέση με τις αποδοχές. Υπήρξε μία μελέτη που είδα που δείχνει ότι ο απλός πολίτης αρχίζει να πιστεύει ότι είναι τελείως άνηση η αμοιβή των στελεχών σε σχέση με τους εργαζομένους. Υπάρχουν χώρες όπως οι Ηνωμένες όπου το μέσο οι μέσες αποδοχές των στελεχών είναι των ανώτατων στελεχών 350 φορές περισσότερες από τον απλό εργαζόμενο στις ίδιες επιχειρήσεις. Επομένως πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να τεθούν κάποια όρια και δεν αρκεί η διαφάνεια. Η ίδια η διαφάνεια που είναι το τρίτο στοιχείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι πάρα πολύ σημαντική. <clears throat> Εδώ υποστηρίζω αυτό που λέει η έκθεση ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε σχέση με τη λογιστική των επιχειρήσεων, τις ε, συναλλαγές μεταξύ συνδεωμένων μερών και την ανταλλαγή πληροφοριών και την διοχέτευση πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερομένους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέγει ο Πρόεδρος η Μόλτ Σκοτ Κέιτο. Καταρχάς θέλω να καλωσορίσω αυτό που είπατε για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της τράπεζας και είναι πολύ θετικό γιατί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ για τη σχετική ανακοίνωση. Για αυτό το ζήτημα τώρα που μας απασχολεί σε αυτό το σημείο της Μέσιας Διάταξης. Χαίρομαι για την ε, νομοδότηση. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό πράγματι να έχουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο τέρκης διακυβέρνησης. Το είδαμε βλέποντας τα διάφορα εταιρικά και δημοσιονομικά σκάνδαλα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας, στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και ως πράσινοι στηρίζουμε τη βελτίωση και περιορισμό των ελλείψεων της εταιρικής κυβέρνησης των εισημένων εταιριών. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επιχειρησιακή διαφάνεια για όλους και να είναι βιώσιμες οι εισηγμένες εταιρείε. Οι προτάσεις κομισιών εστιάζουν στους μετόχους βέβαια. Εμείς στηρίζουμε την άποψη του εισηγητή να συμπεριληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να περιλαμβάνονται δηλαδή οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι και η τοπική κοινωνία, με, τους οποίους, ε, με τα μέλη της οποίας έχει σχέση η εταιρεία. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ενεργό συμμετοχή και σεβασμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων που ε, επηρεάζονται από τη στρατηγική της εταιρείας. Από την πράσινη σκοπιά και γιατί θέλουμε να υπάρξει μακροπρόθεσμη εστίαση, η διαφάνεια των εταιρικών αποφάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει και ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή αναφορέα σχετικέ. Θα πρέπει και τα λεγόμενα δεσμευμένα στοιχεία, ε, περιουσιακά στοιχεία, stranded assets να ε, ερευνώνται. Πού είναι αυτά τα στοιχεία. Και βέβαια και οι εκπομπές οξυδίου του άνθρακα είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Επίσης, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη εξουσία σε αυτούς που λαμβάνουν συντάξεις Μήπως πρέπει επίσης να δημιουργηθεί να αντιπροσωπευτική, ε, αντιπροσωπευτικές δομές ή αντιπροσωπευτικοί φορείς αυτών των εμπλεκομένων φορέων. Τώρα, συγκεκριμένες τροπολογίες. Εμείς θα εστιάσουμε στα εξής στις δικές μας τροπολογίες. Στο ένα βελτίωση του διαλόγου. Το στηρίζουμε. Αλλά θα θέλαμε, για να μην υπάρχουν ε, πιθανές εντάσεις ή να υπάρχουν εταιρικά μοντέλα επιχείρησης για να υπάρχει συνεργασία. Το μοντέλο του Τζον Lewis πέτυχε επειδή πρόσφατα φάνηκε ότι μπορεί να αντέξει και τις δύσκολες συνδίκες της αγοράς. Θέλουμε και τη συμμετοχή των εργαζομένων, να υπάρχει προχωρητική εκπροσώπηση του στα Σίγμα Και θα πρέπει να υπάρχει διάλογος ε, με τη διοίκηση της εταιρείας για να υπάρχει διαφάνεια και να λαμβάνονται υπόψη στις εταιρικέ αποφάσεις όλοι οι φορείς. Δεύτερο σημείο, διαφάνεια. Καλή είναι η σχετική δέσμευση, αλλά θα πρέπει οι διευθυντέ και άλλοι σημαντικοί φορείς να παίρνουν πραγματικά την ευθύνη των αποφάσεών τους. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει ε, για τους λογιστές εξαιρετικούς ελεγκτές ένα επιπλέον ε, για να μπορούν να τους ελέγχουν καλύτερα και ενδεχομένω και επιβολή προστήμων ή κυρώσεων ή πάυση από τις θέσεις για τους επιλεξούς συμβούλους. Για τις αποδοχές συμφωνώ και πράγματι θα πρέπει να ελέγχουν οι μέτοχοι την αναλογία των αποδοχών των ε, εργαζομένων ε, και των διοικητικών στελεχών. Είναι καλή η βάση του σχεδίου γνωμοδότηση για συμβιβασμό. Θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή και του σκιώδε των άλλων ομάδων. Ευχαριστώ. Thank you to the Ευχαριστώ τους σκιώδεις και τους εκπροσώπους των σκιωδών θα δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή για τις τελικές του παρατηρήσεις για να κλείσει η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα εγώ είμαι δεκτικός για να προχωρήσει ο διάλογος και να μπορέσουμε να βρούμε κοινέ θέσει και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ευρεία βάση στήριξης της έκθεσης αυτής. Υπάρχει εδώ ένα σημείο που έχει σημασία και έχει άμεση σχέση με τον ρόλο των μετόχων. Ε, σας ευχαριστώ καταρχάς για τις προτάσεις σας. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση και θα τα καταφέρουμε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Η προθεσμία κατάθεσης είναι η 6η Ιανουαρίου 12η μεσημβρινή εξέταση των τροπολογιών θα γίνει την 26 Ιανουαρίου. Η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ προβλέπεται για την 31η Φεβρουαρίου, 21η συγγνώμη, Φεβρουαρίου. Η ψηφοφορία στην Αρμόδια Επιτροπή θα γίνει την 24η Μαρτίου και ε, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια μετά το Μάρτιο. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ετήσια έκθεση. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή Ουρτασούν από πλευρά των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω <clears throat> ξεκινώντας να ευχαριστήσω για την εκπόνηση αυτού του εγγράφου που έχετε ενώπιόν σας από... Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους εκπροσώπους της ομάδος επενδυτών και είναι κάποιοι από αυτούς εδώ παρόντες. Είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε την Τράπεζα Επενδύσεων τον Νοέμβριο και είδαμε πως έχουν τροποποιηθεί τα πράγματα μετά από την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δεύτερη ευχαριστία μου, πέραν της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, απευθύνεται βέβαια στους κοιόδησης οι οποίοι αντιμετώπισαν και αυτοί το θέμα αυτό, με του οποίους είχα τη δυνατότητα να κάνουμε συζητήσει <clears throat> και νομίζω ότι υπήρξε μια θετική α, θέληση από όλου να μπορούμε να έχουμε μια συνενετικού χαρακτήρα έκθεση. Και φυσικά εδώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πλαίσιο της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο μελλοντικό σχέδιο επενδύσεων που έχει παρουσιαστεί στην προηγούμενη Ολομέλεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είναι στόχος της τρέχουσας έκθεσης να κάνει μια συνελική αξιολόγηση του σχεδίου Juncker, γιατί ξέρετε όλοι ότι αυτό θα γίνει από μια χωριστή έκθεση η οποία θα αναφέρεται αποκλειστικά στο θέμα αυτό. Φυσικά όμως <clears throat> είναι υποχρέωση του εισηγητού και των σκιωδών να αναλύσουν τον ρόλο που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και νομίζω ότι υπάρχει μια συνένεση αυξανόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τη στιγμή που υπάρχει μείωση των επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη χρειαζόμαστε μια πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ώστε να μπορέσει να μειωθεί το χάσμα επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο λοιπόν έκθεσης που έχετε ενώπιόν σας παρουσιάστηκε στις 20 του μηνός, δηλαδή πριν του Νοεμβρίου, δηλαδή πριν από την ανακοίνωση του σχεδίου επενδύσεων Juncker. Κάποια σημεία λοιπόν, όπως το σημείο 3, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν στην έκθεση αυτή. Αυτό είναι κάτι που συζητήσαμε μεταξύ των σκιωδών εισηγητών την προηγούμενη εβδομάδα και φυσικά πολλά στοιχεία μπορούν να καλυφθούν και από τη διαδικασία κατάθεσης τροπολογιών ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα συγκεκριμένα στοιχεία του σχεδίου Juncker. Η έκθεση είναι οργανωμένη σε τμήματα. Το πρώτο τμήμα για τις επενδύσεις, το δεύτερο για τις, ε, τις ομολογίες που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση των επενδύσεων, τα μέσα επιμερισμού κινδύνου επίσης. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία είναι αποτελέσματα της ε, Συνόδου του Παρισιού πέρσι, επίσης για τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια και τέλος για τον εξωτερικό αντίκτυπο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μπορούμε να σταθούμε σε κάποιες λεπτομέρειες για το πρώτο μπλοκ της επενδύσεις. Ξέρουμε όλοι ότι έχουν μειωθεί κατά 18% από το 2007 οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης έχει μειωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η <clears throat> οποία υπολογίζεται σε περίπου 35%. Αυτό ήταν ένα σημαντικό θέμα το οποίο τον τόνισαν πολλοί σκιώδεις εισηγητές ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό με τη μείωση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να το εξάρουμε. Σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις επενδύσεις, τονίζει η έκθεση ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μια οικονομική ανάκαμψη γιατί υπάρχουν προβλήματα ήδη με την ε, στρατηγική του 2020 σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την καταπολέμηση της ένδυας. Η έκθεση λοιπόν κάνει και μια ε, προτροπή στην ενίσχυση της ικανότητας δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην αύξηση των στοιχείων ενεργητικού της κτλ. Τονίζει επίσης η έκθεση και το γεγονός ότι υπήρξε υποχρησιμοποίηση των δυνατοτήτων δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων παρά το γεγονός ότι ενισχύθηκε το κεφάλαιο αυτής της τράπεζας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ. Τέλος για τα θέματα επενδύσεων. Αν λάβουμε υπόψη το υψηλό επίπεδο ανεργίας το οποίο σοβεί στα περισσότερα μέλη της κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητούμε από την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων να αντιμετωπίσει τα θέματα ανθρωπίνου κεφαλαίου και απασχόλησης. Το δεύτερο τμήμα που είναι η ορθιμερισμός κινδύνου και τα ομόλογα έργων κάνουμε κάποια κριτική για τα μέσα επιμερισμού κινδύνου και σε σχέση με τις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν για τη χρήση αυτών των μέσων και κάνουμε και μια αξιολόγηση των νέων εργαλείων που έχουν τεθεί σε λειτουργία τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένα τα ομόλογα έργων, project bonds, που είναι πολύ σημαντικά λοιπόν νέα στοιχεία και που βρίσκονται ακόμα στη φάση, στην πιλωτική, στη φάση εκκίνησης. Κάνουμε λοιπόν μια κριτική ανάγνωση όλων αυτών των εργαλείων, συγκεκριμένα για το σχέδιο Κάστορ, το έργο Κάστορ, και κάνουμε μια εντελεχή ανάλυση για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση αυτή και τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Στο τρίτο μπλοκ που έχει να κάνει με την ενέργεια και το κλίμα, ε, ασχολούμαστε με την θέληση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να ακολουθήσει μια νέα πολιτική σε επίπεδο ενέργειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζητούμε να μειωθεί η επένδυση σε ενεργειακή παραγωγή που χρησιμοποιεί άνθρακα. Τονίσουμε την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν καλύτερα τα σχέδια ανανεώσιμης ενέργειας και φυσικά και να υπάρχει και μεγαλύτερη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ζητούμε επίσης να υπάρξει μια σταδιακή απόσυρση <clears throat> των ε, χρηματοδοτήσεων για συμβατικές ενέργειες. Σε ό,τι αφορά τώρα τη κυβέρνηση, διαφανεία και λογοδοσία, που είναι ένα τμήμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε τονίσει την ανάγκη μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κάνουμε κάποιε εκτιμήσει, οι οποίε μου φαίνονται πολύ σημαντικέ. Κάνουμε μία έκκληση για καλύτερο μηχανισμό έγερσης αντιρρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει λειτουργήσει σε ό,τι αφορά την υποδοχή παραπώνων ή ε, ενστάσεων από τους πολίτες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε βέβαια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δεχτεί αυτό το μηχανισμό υποβολής παραπώνων. Τονίζουμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία με τους πολίτες και την κοινή γνώμη. Η έκθεση επίσης <clears throat> αντιμετωπίζει τα θέματα των ε, διαμεσολαβητών στο χρηματοπιστωτικό χώρο. Ζητούμε να περιοριστεί η συνεργασία με αυτούς, να μην συνεργαζόμαστε με σκιώδεις ή αδιαφανείς ε, οντότητες στο χρηματοπιστωτικό τομέα και χαιρόμαστε για το γεγονό ότι δημιουργείται ένα δημόσιο μητρό εγγράφων. Και τέλος, και κλείνω εδώ πέρα, υπάρχει το μπλοκ για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ζητούμε να υπάρξει μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των ε, δράσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ληφθεί υπόψη το κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο των χώρων όπου γίνεται αυτή η επένδυση και θέλουμε να υπάρξει ένα, ένα μέσο καταμέτρησης των αποτελεσμάτων των ε, χρηματοδοτήσεων αυτών που μπορεί να μας βοηθήσει στο μέλλον. Και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι δημοσιεύονται οι πληροφορίες για την <clears throat> περάτωση των ε, προγραμμάτων και των σχεδίων και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό και επομένως ζητούμε να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό. Κλείνω λοιπόν κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι μια έκθεση η οποία αντιμετωπίζει τα θέματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε διάφορους τομείς όλο το πακέτο των επενδύσεων είναι πολύ, το νέο πακέτο επενδύσεων είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή της τράπεζας στα θέματα των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητη να υπάρξει μια αξιολόγηση κατά τομή των εργαλείων και να τονίσουμε τη δημοκρατία και την ε, διαφάνεια. Και είμαι στη διάθεση των σκιωδών για τα σχόλιά τους και για τη μελλοντική εργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μάλλον Μουρεσάν για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας να ευχαριστήσω τον εισηγητή με τον οποίο μπορέσαμε να συνεργαστούμε με καποφόρο τρόπο στα πλαίσια της διαδικασίας σύνταξης της έκθεσης και ελπίζω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί του και με τους κοιόδης των υπολείπων πολιτικών ομάδων μέχρι την τελική υιοθέτηση της έκθεσης στην Ολομέλεια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει πράγματι αποκτήσει μεγάλη σημασία στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης για να βοηθήσει να ξεπεραστεί η συγκεκριμένη κρίση σε σχέση με τη στήριξη των δημοσίων επενδύσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία και την αποκατάσταση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτό υπογραμμίστηκε και από τον ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Επενδυτική αυτή τράπεζα στα πλαίσια του πακέτου του επενδυτικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ασχοληθούμε βέβαια με αυτό το πακέτο το επενδυτικό σε μια άλλη έκθεση και δεν θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό. Να πω παρόλα αυτά όμως ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε το πακέτο αυτό το επενδυτικό να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να φέρει εις πέρα στην αποστολή της και θα επιτρέψει επίσης στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ολοκληρώσει την αποστολή του. Σχετικά τώρα με το πακέτο των 300 δις και τις επιπτώσεις του στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να δούμε αν μπορεί να υπάρξει ένας νέος ρόλος για την τράπεζα αυτή, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και στην ανάγκη περαιτέρω προσωπικού για να φέρει πέρα στις νέες αποστολές της. Έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μην έχει προβλήματα έλλειψης προσωπικού. Είναι γεγονός ότι έχει αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις της το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά 37% κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της αύξησης των κεφαλαίων της τράπεζας την οποία και εμείς στηρίξαμε. Η ομάδα μας θεωρεί ότι έχει παίξει λοιπόν συνολικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ένα θετικό ρόλο στην στήριξη ε, των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και νομίζω ότι η έκθεση μετά από κάποιες αλλαγές που έγιναν στην αρχή ξεκινάει με κάποιες παρατηρήσεις και κριτικές προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε σχέση με τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι σίγουρα η μοναδική υπεύθυνη για τη μείωση των επενδύσεων. Και ξεκινώντας με τέτοιο αρνητικό τρόπο την έκθεση νομίζουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο δείχνει τις προσπάθειες της τράπεζας και τις βελτιώσεις των τελευταίων χρόνων, όπου έπαιξε ένα θετικό ρόλο η τράπεζα για την αύξηση των επενδύσεων και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κάποια επιπλέον σημεία για τα διαφορετικά τμήματα της παρουσίασης που έγινε από τον εισηγητή. Ο εισηγητής πάρα πολύ σωστά μίλησε για τις δύσκολες συνθήκες για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Όλοι πιστεύουμε ότι οι μικρομεσαίες δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη και οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι οι καλύτερες στήριξε 130.000 περίπου βέβαια τα τελευταία χρόνια και αυτή η χρηματοδότηση έφτασε τα 21 δις. Είναι αρκετά σημαντικά αυτά σαν ποσά και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ξεχωριστή, ε, ένα ξεχωριστό τμήμα για τις μικρομεσαίες στην έκθεση, στην ετήσια έκθεση. Θα πρέπει να διαβρινθεί λοιπόν και να στηριχθεί η επένδυση προς τις μικρομεσές ε, και μέσω των, ε, μέσων μικροεπενδύσεων, μικροχρηματοδότηση συγγνώμη, ιδιαίτερα τη στήριξη καινοτόμων μικρομεσαίων και αυτό με οδηγεί στο επόμενο σημείο. Η καινοτομία, η έρευνα και οι υποδομές είναι επίσης τομείς τους οποίους θα θέλαμε να υπογραμμιστούν καλύτερα. Ναι λοιπόν στις μικρομεσαίες, ναι στην έρευνα, ναι στην καινοτομία, ναι στις υποδομές. Ε, όλα αυτά θα καταστήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία ανταγωνιστικότερη και ελκυστικότερη για τους επενδυτές. Αναγνωρίζω ε, θετικά εννοώ τον ρόλο της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας στη χρηματοδότηση των λεγόμενων καθαρών προγραμμάτων και θα πρέπει να συνεχιστεί η τάση αυτή. Έχω κάποιες ανησυχίες βέβαια γιατί μόνο ένα από αυτά τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκε με δημόσια ομόλογα περιλαμβάνεται στην έκθεση. Και θα πρέπει εμείς με τον εισηγητή να δούμε αν θα αναφέρουμε όλα τα προγράμματα ή μόνο ένα από αυτά ή κανένα από αυτά. Νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσουμε καλύτερα. Ε, για τον ρόλο της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και εδώ η τράπεζα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να μην αγνοούμε ότι πρόκειται για μια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όχι γενικότερα για το θέμα της αποδοτικότητας της ενέργειας και για τις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών. Εμείς θα πρέπει να ελέγξουμε αν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εντάσσεται στους στόχους τους γενικότερους που έχουμε τώρα για τα ομόλογα έργου. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε και το θέμα της ε, Investment and uh, the mutualization of debt in whatever form is no replacement for um, uh, economic reforms, for structural reforms, for measures which lead to... Θέματα του επιμερισμού του χρέους και είναι θέματα τα οποία θα στηρίξουν γενικότερα τις πολιτικές μας και θα βοηθήσουν και μια σωστότερη δημοσιονομική πολιτική. Για τα θέματα της διαφάνειας, εδώ συμφωνώ με την έκκληση του εισηγητή, ο οποίος ζητά να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και τις προσπάθειες που έχει ήδη κάνει η τράπεζα ε, για τα θέματα αυτά τα τελευταία χρόνια. Um, um, είναι θέματα λοιπόν τα οποία έχουν ε, εξεταστεί και στα πλαίσια της έκθεσης για τα θέματα της διαφάνειας γενικότερα και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στις ε, στους κύκλους εργασίας τους οποίους έχει αυτή τη στιγμή η, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και κάτι το οποίο με ενδιαφέρει επίσης είναι και η εμπλοκή της τράπεζας στην Ανατολική Γειτονία, Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία που ακολουθούν τον Ευρωπαϊκό δρόμο και έχουν ως εκ τούτου σημαντικό ρόλο να παίξουν για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα βέβαια οι σκιώδεις να μην μακρηγορήσουν τόσο πολύ. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους ε, των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, ο Ρίτσαρτ Κόρπετ, μέρους σκιώδους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ο σκιώδης διοικητής, ο κύριος Μπαγιέ, είναι ένας από τους οποίους ε, καθυστερεί λόγω των προβλημάτων στην κίνηση σήμερα. Ευτυχώς όμως. Μου έδωσε τις σημειώσεις του. Αλλά βάλτε ακουστικά γιατί θα τα διαβάσω και είναι στα γαλλικά τα σχόλια. Καταρχάς λοιπόν ε, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ο κύριος Μπαγί λοιπόν ε, θεωρεί ότι έχετε κάνει καλή δουλειά και είναι καλή βάση αυτό το έγγραφο. Κάνουμε λοιπόν έναν πολύ σωστό προβληματισμό για την, ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή μάλλον, Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει τι δυνατότητε αυτή τη τράπεζα να τι εντάξουμε στο διεπτόν καλύτερα στο επενδυτικό σχέδιο που πλέον δρομολόγησε ο κ. Γιούγκερ. Τα ομόλογα έργων θα μπορούσαν να, δώσουν ε, μια νέα πνοή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα νέο δυναμικό. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε μια γρήγορη αξιολόγηση των υλοποιούμενων έργων. Και βέβαια πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα ταμεία, όλα τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας ε, του παρόντος, το ποσοστό χρήσης ανέρχεται στα 2 τρίτα των διαθέσιμων κονδυλίων μόνο. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουμε όλους τους δυνατούς μοχλούς για να ασκήσουμε τις πιέσεις για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Και Κατά τούτο και για να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσο θα το περισσότερο θα πρέπει να υπάρξει μια κατάλληλη διαδικασία διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους φορείς. Αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να βελτιώσει και την αξιολόγηση των έργων στην οποία προβαίνει, λαμβάνοντα υπόψη και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Είναι μια ε, διαδικασία από κάτω προς τα πάνω και τη γνωρίζουμε ήδη σε ορισμένες χώρες από τα διαρθρωτικά ταμεία. Σε ό,τι αφορά τώρα τους στόχους των υποστηριζόμενων σχεδίων και έργων. Είναι επίγον μεταξύ άλλων να χρηματοδοτηθούν πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ε, μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, ε, ώστε να μπορέσουμε να σεβαστούμε τις προτεραιότητες που έχουμε σε ό,τι αφορά τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου των εκπομπών αυτών των αερίων. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαφάνεια και την χρηστή διακυβέρνηση, είναι σημαντικό ότι η ΕΤΕΠ δεν θα πρέπει να συνεργάζεται με χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, ε, όμως σε δικαιοδοσίες με τις οποίες δεν υπάρχει συνεργασία. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε το Λουξεμβούργο, το Μαυρίκιο και άλλα παραδείγματα τέτοια μη συνεργάσιμων ε, χωρών. Η καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων πρέπει να είναι μια προτεραιότητα για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο και για τα θεσμικά όνα της Ένωσης, μεταξύ των οποίων και για την ΕΤΕΠ που θα πρέπει να είναι πρότυπο για υπόδειγμα στον τομέα αυτό. Άλλο, η ΕΤΕΠΑ θα πρέπει να καταφεύγει σε κάποιους ιδιωτικούς συμβούλους ε, για την ε, αξιολόγηση κάποιων στοιχείων. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα για να βοηθηθούν περισσότερο οι ΜΜΕ, που θα μπορούσαν να ορίζουν οι ίδιες κριτήρια και την διαφανή μεθοδολογία για την ανάλυση των κινδύνων για να μην περνούν πλέον μέσα από ιδιωτικές εταιρείε για το σκοπό αυτό. Τέλος, ό,τι αφορά την εξωτερική βοήθεια. Αυτό το σημείο λοιπόν ήταν η η αξιολόγηση ε, και για τα εξωτερικά συμφωνούμε με τον εισηγητή. Thank you, Richard. Next speaker for the EC. Ευχαριστώ, Richard ο Στάνισλαβ Ζοκ από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όπως σου είπε ο Πρόεδρος θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω. Ο εισηγητής ήταν από την αρχή πολύ ανοιχτός σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου με τους σκιώδεις εισηγητές, ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια την οποία έχει ήδη καταβάλει ο εισηγητής. Η έκθεση προχωρεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά την άποψή μου και μπορώ να, συνεχίσω, μπορώ να συμφωνήσω με την αναφορά στο σχέδιο Juncker, αλλά τα 300 δισεκατομμύρια έχουν ήδη εγκριθεί και δεν είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος για να κάνουμε μια συζήτηση. Τώρα, για το κείμενο σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των σχεδίων, εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να γίνεται πλήρως και με δημόσια διαβούλευση, εάν έχει αντίκτυπο σε κοινωνικό επίπεδο και στις τοπικές κοινότητες. Επίση είναι σημαντικό να αναλύονται και τα οικονομικά ωφέλη σε επίπεδο ανάπτυξης και απασχόλησης που θα προέρθουν από ένα σχέδιο, ιδίω σε περιοχές με υψηλή ανεργία. Επίσης αναφέρεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα στα σχέδια ο εισηγητής και εδώ θα ήθελα να αναφέρεται και περισσότερο το οικονομικό όφελος και όχι μόνο η ενεργειακή απόδοση. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν πολλές μνήες αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Νομίζω το 2013 έφτασε στα 30% και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Η υποστήριξη των μικρομεσαίων είναι πολύ σημαντική για να υπάρχει δημιουργία θέσεων επί απασχόλησης στις τοπικές κοινότητες. Η έκθεση αυτή λοιπόν θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο σε αυτό τον τομέα. Το 2013 για πρώτη φορά ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις μικροχρηματοδοτικού χαρακτήρα στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε ίσως περισσότερο και τέλος εγώ υποστηρίζω τον εισηγητή μας θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει σχέδια τα οποία εστιάζουν περισσότερο στην ενεργειακή απόδοση αλλά δεν θα πρέπει να προκαταλάβουμε την επιλογή των προγραμμάτων που θα πρέπει να ε, καταργηθούν εν καιρό. Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω το κεφάλαιο 20, την παράγραφο 20 του κειμένου ως έχει. Ευχαριστώ. Thank you. for... Ευχαριστώ για την ομάδα της Άλντε, ο κύριος Γέτζεκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσής του και για την θέλησή του να επιτύχει μια ευρεία συνένεση με την δική του ιδιαίτερα θετική προσέγγιση. Υπάρχουν πολλά λοιπόν ισχυρά στοιχεία στην έκθεση που θα ήθελα να επικροτήσω, αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που είπε και ο προηγούμενος ομιλητής. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην έκθεσή του, αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Νομίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι, είναι κέριο στοιχείο της ευμάρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη επένδυση στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004, ιδίως για σχέδια που έχουν να κάνουν με ενεργειακή απόδοση. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν γενικά επωφελές και θα βοηθούσε να μπορέσουμε να περάσουμε από την κατανάλωση άνθρακος στην παραγωγή ενέργειας σε μια πιο ε, ε, χαμηλού αποτυπώματος άνθρακος ε, οικονομία. Η Ευρώπη βρίσκεται στο προσκήνιο, είναι πρωτοπόρος στα θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και ως εκ τούτου αυτό θα πρέπει να χαιρετιστεί. Παράλληλα όμως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν άλλοι τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση στερεί εναντί των ανταγωνιστών της, παγκοσχάρη χάρη, στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για το σχέδιο Juncker νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να εστιάσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όχι στο συγκεκριμένο αυτό σχέδιο. Γιατί αυτό θα είναι το αντικείμενο άλλων εκθέσεων. Γενικά είναι πολύ καλό σημείο κίνηση αυτή η έκθεση και είμαι έτοιμος να συζητήσω περαιτέρω με τον εισηγητή και να καταθέσω σχετικές τοπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο για την ΚΟΕ. Ο κύριος Παπαδημούλης, όχι, η Μαρίζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Δυστυχώς όπως καταλαβαίνετε με τις απεργίες δεν μπόρεσε να έρθει ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Εγώ θα προσπαθήσω λοιπόν να τον εκπροσωπήσω εδώ όσο αυτό είναι εφικτό. θα ήθελα να αναφέρω αυτά τα οποία μου έχει αποστείλει υπομορφή σημειώματος ο κύριος ε, Παπαδημούλης. Κάποια από αυτά τα στοιχεία αναφέρθηκαν και από τον εισηγητή στην αρχική του παρέμβαση, αλλά εγώ θα σταθώ στα σημεία αυτά τα οποία ε, μου είδε ο κ. Παπαδημούλης και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή ο Δημήτρης. Πιστεύει ότι το σχέδιο έκθεση είναι μια πολύ καλή προσπάθεια και μια πολύ καλή βάση εργασίας για την μελλοντική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα κέρια θέματα. αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το εξής. Τα θέματα της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Και εδώ ο Δημήτρης θα ήθελε να τονίσει ποια είναι τα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα με τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η επιλογή των σχεδίων, η καταλληλότητα των σχεδίων και τα θέματα συναλλαγών με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές. Ζητά να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιότητα σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλει να γύρει ο κ. Παπαδημούλης είναι η αλλαγή νοοτροπίας της τράπεζας. Είναι ε, μια νοοτροπία τραπεζικού χαρακτήρα η οποία δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της ε, ευρείας κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. Πολλές φορές η αποδοτικότητα σε <clears throat> χρηματοπιστωτικό επίπεδο υπερτερεί τις ανάγκες να υποστηριχθούν κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι. Επομένως, θα πρέπει να μην περιορίστε στη διατήρηση του τριπλού αλφα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μπορεί αυτό να αποτελέσει ένα πρόσκομα για επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν την πραγματική οικονομία και πάλι στον δρόμο της ανάκαμψης και της απασχόλησης. Ένα τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με την μεγαλύτερη ικανότητα δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλείται να παίξει ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο για τις χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα ή που είναι σε διαδικασία εξυγίανσης. Μπορεί να υποστηρίξει στην ανάκαμψη, προωθώντας τις επενδύσεις, ενισχύοντας την απασχόληση και μια τέταρτη ανησυχία αφορά την επανεκτίμηση της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα έργο και εδώ η συνάδελφος ε, ε, είπε πάρα πολλά και με τα οποία συμφωνούμε, αλλά θα διαβάσω τις σημειώσεις μου. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό είναι ε, το κατάλληλο μέσο τα ομόλογα έργου για αυτού του είδους τις επενδύσεις. Εμείς έχουμε επιφυλάξει σχετικά με τα PPIs. είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εμπλακούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και θα πρέπει επίσης να δούμε αν τα προγράμματα υποδομών θα χρηματοδοτηθούν από το δημόσιο χρήμα παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις και απαιτήσεις των πολιτών. Έχει σημασία λοιπόν να προσπαθήσουμε να προσέξουμε ε, τα προγράμματα αυτά αποφεύγοντας ψευδοπρογράμματα και ασύμετρα προγράμματα. Ο Δημήτρης δίνει και κάποια παραδείγματα στα οποία υπήρξαν αναφορές το πρόγραμμα Κάστορ στην Ισπανία ή το πρόγραμμα Πασάντε που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτού του είδους τις αναλύσεις. Μια πέμπτη ανησυχία του Δημήτρη αφορά την α, μακροοικονομική προσθετικότητα για τις πρωτοβουλίες τις επενδυτικές. Δεν θα πρέπει να συνδέονται με τα προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Δεν πρέπει να είναι η πρόοδος ενός τέτοιου προγράμματος προϋπόθεση για τα επενδυτικά αυτά σχέδια. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε στην ενίσχυση της έκθεσης με τις δικές μας τροπολογίες και να ευχαριστήσουμε και τον εισήγητη. Ευχαριστώ λέω Γκουαλτιέρη, Γκουτσάνη. Η συνάδελφος Πούλτο δεν είναι παρούσα, λέει ο κύριος Βάλλη. Ασχολήθηκα με το ίδιο θέμα σαν συντονιστής για την πολιτική μου ομάδα και στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ιδιαίτερα για τα ομόλογα έργο. Ανησυχούμε ιδιαίτερως γι' αυτά Ήδη στο πρόγραμμα του 2012 είδαμε ότι τέτοιου είδους προγράμματα μερικές φορές οδηγήθησαν σε πλήρη αποτυχία. Είδαμε τι έγινε με το Πατσάντε στο Μέστρε, είδαμε το Κάστορ στο Μέστρε, οι τοπικές αρχές είπαν ότι υπάρχει ισχώρηση του οργανωμένου εγκλήματος στους διαγωνισμούς και στις προμήθειες και γιατί δυστυχώς όπου υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα έργα υπάρχουν και τα πλοκάμια του οργανωμένου εγκλήματος για να κλέψουν το δημόσιο χρήμα, όπως είπε και συνάδελφος από την Άλντε. Το θέμα είναι λοιπόν από τα προγράμματα αυτά να ωφεληθούν οι τοπικές οικονομίες και σε επίπεδο απασχόλησης, γιατί αλλιώς οι πόροι θα πρέπει καλύτερα να κατευθυνθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί θα είναι πιο αποδοτικές. Και οι εταιρείε αυτές οι μικρομεσαίες ίσως δίνουν περισσότερες εγγυήσεις σε επίπεδο απασχόλησης από ότι ένα πολύ μεγάλο δημόσιο έργο. Ένα πολύ μεγάλο δημόσιο έργο, όπως είπα, προσελκύει το οργανωμένο έγκλημα. Ελπίζω ότι το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει ο Γιούνκερ και για την Ιταλία, για την οποία υποτίθονται απευθύνονται 87 δις, δεν θα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα έργα όπως το ή το Οτάβο κτλ. Ευχαριστώ. Το Catch πλέον. Άνεμανς. Μη εγγεγραμμένος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Υπάρχει μια λογική πίσω από τις προτάσεις αυτές, όπως ακούστηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές. Η επιλογή των πιστώσεων, των προορισμών μάλλον των πιστώσεων, γίνεται ουσιαστικά εκτός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει οδηγήσει την ευρωπαϊκή οικονομία στο μηδέν. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική αυτή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να παρεμβαίνει μεν, αλλά εξισοπηρητικά. Γιατί στην ουσία σε σχέση με τις σημαντικές επενδύσεις η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αποχωρήσει. Θα πρέπει να λειτουργήσει με συμπληρωματικό τρόπο. Είναι ένα μέσο το οποίο τροφοδοτείται από το χρήμα του φορολογούμενου, να μην το ξεχνάμε και είναι και ένα μέσο το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχει ο κόσμος απέναντι στη ζώνη ευρώ και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχει οδηγήσει σε μηδενική ανάκαμψη. Υπάρχει λοιπόν ένα παράδοξο εδώ, μια αντίθεση. Μιλάμε για προτάσεις οι οποίες ε, δεν σέβονται την σύμβαση της Βασιλείας, και δεν μπορούν έτσι τα πιστοτικά ιδρύματα να λειτουργήσουν σωστά και να ξαναβάλουν την οικονομία σε λειτουργία. Θέλουμε επίσης να υπογραμμίσουμε και το θέμα της αηφορίας και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Θυμίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ιδιωτών επενδυτών έχει αποχωρήσει ουσιαστικά και δεν θέλει να επενδύει στην Ευρώπη μακροπρόθεσμα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και ένα τελευταίο παράδοξο είναι αυτό το οποίο λέτε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι θα πρέπει να λειτουργήσει σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο και να καλύψει τις ανάγκες ε, ε, που έχουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο πρέπει να χαρακτηρίσει με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο μέλλον, αλλά αυτό δεν αναιρεί τα σημαντικά προβλήματα τα οποία δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει από μόνη της αυτή η τράπεζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι είναι πολλά ενδιαφέροντα σημεία που αναφέρονται στην έκθεση αυτή σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ιδίως αυτά που έχουν να κάνουν με μικροχρηματοδοτήσεις ή με την ε, συμπερίληψη σε κοινωνικό επίπεδο, την επένδυση το προς όφελος των νέων. Όλα αυτά είναι λοιπόν πολύ θετικά. Ξέρω ότι οι και άλλοι έχουν αναφερθεί στο πακέτο Ιούνκερ και τον κέριο ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θέλω εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό ότι η ομάδα που θα δημιουργηθεί για την επιλογή των πρόων των σχεδίων δεν θα επιλέξει μονάχα, να μην επιλέξει μονάχα τα εύκολα σχέδια. Δεν πρέπει εμείς να εστιάσουμε σε σχέδια τα οποία ήδη υπάρχουν, έχουν ήδη αξιολογηθεί. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το πακέτο αυτό επενδύσεων θα είναι προσβάσιμο σε όλους. Είναι απαραίτητη λοιπόν <clears throat> η διαφάνεια για να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία και να έχουμε και την ευκαιρία να έχουμε μια πλήρη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα πρέπει να τροποποιηθεί και να είναι πιο κέριος στο μέλλον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και ο Πρόεδρος, η Κάθριν Στάιλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους σκιώδες για τη συμβολή τους. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση η οποία έχει λάβει η χώρα και τονίζει και πάλι τη σημασία του ρόλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα ήταν χρήσιμο να μας δώσει ένα κατάλογο των σχεδίων που χρηματοδοτούνται για κάθε συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης. Γιατί πολλές φορές όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι γνωστά στον πληθυσμό. Ίσως μπορεί να το αναλάβει αυτό η εισηγήτης, να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα σχέδια τα οποία χωρίς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί. Και ιδίω όταν πρόκειται για τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λέει η έκθεση, ότι προβλέπονται 21, είναι 21,9 δισεκατομμύρια που πήγαν σε χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Αν είχαμε όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να πάμε στις εκλογικές μας περιφέρειες και να εξηγήσουμε πώς τις βοήθησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης, στην Διαχειριστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπάρχει μονάχα μία γυναίκα και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο εγώ θέλω να είμαι λίγο πιο κριτική, γιατί εμείς πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία των γυναικών και εγώ βλέπω να είναι απογοητευτικό να μην υπάρχει μια τέτοια μνήα από τον εισηγητή αυτού του σημείου. Και επίσης το 1 τρίτο της ε, χρηματοδότησης που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή <clears throat> είναι κάτι το οποίο πρέπει να το χαιρετήσουμε ιδιαίτερα. Αλλά και πάλι να τονίσω το θέμα των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπεντ Λούκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα θέλω να προσθέσω για αυτή την έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να προσπαθήσει να είναι πιο συγκεκριμένη στις παρεμβάσεις της σε περιφερειακό επίπεδο να δει πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα χρηματοδοτικά κενά τα οποία είναι πολύ άνισα κατανεμημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και στην Ευρωζώνη. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εστιάζει την προσοχή της όπου υπάρχει το μεγαλύτερο χάσμα επενδύσεων και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την σχέση δημοσίων επενδύσεων και το ρόλο τους στη δημιουργία υποδομών και της ιδιωτικής επένδυσης σε κάθε χώρα. Εκεί θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένη λοιπόν η κατάσταση, να αντιμετωπίζεται ε, διαφοροποιημένα και να βλέπει που πράγματι υπάρχει μια έλλειψη επαρκών υποδομών στα θέματα ε, υποδομών, αν είναι το πρόβλημα δηλαδή η έλλειψη υποδομών ή αν υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να είναι λοιπόν καλύτερα στόχοθετημένη η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ό,τι αφορά την πρόθεση των επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Θα ακούσουμε την ίδια την τράπεζα τώρα. Κύριο Κνάπεν, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας της ευρωπαικης τραπεζας επενδυσεων σε οτι αφορα την πρόοδο των επενδυσεων ευχαριστω ευχαριστω λεει επενδύσεων της Βρυξέλλες. επενδυσεων της Βεξέλλες. ευχαριστω προεδρε Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και ιδιαίτερα τον κύριο Ούρτασούν για τις προσπάθειες τις οποίες έκανε. Έχει σημασία φυσικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί σε αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να σας πω όμως ότι αυτό λειτουργεί και αμφίδρομα για μας, πως που εργαζόμεθα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει, ε, είναι, μεγάλη, είναι πολύ σημαντικό το να μας ελέγχει με δημοκρατικό τρόπο το Κοινοβούλιο. Και είδα ότι και στο παρελθόν οι παρατηρήσεις σας έχουν δημιουργήσει θα έλεγα έχουν πλέον μια μόνιμη παρουσία στα διάφορα τμήματα της τράπεζας και λαμβάνονται συστηματικά υπόψη. Λοιπόν, θα ασχοληθώ με κάποια επιμέρους θέματα τα οποία έχουν τεθεί γενικότερα από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Πρώτον, η συζήτηση αυτή έρχεται σε την κατάλληλη στιγμή Βρισκόμαστε στο μέσο μιας νέας επενδυτικής προσπάθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ε, παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε όλοι υπόψη. Να δούμε ότι η αύξηση κεφαλαίου την οποία πήραμε, κερδίσαμε πριν δύο χρόνια, μας επέτρεψε να κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις σε προγράμματα που έφτασαν στα τρία χρόνια τα 180 δις. Τώρα είμαστε στο τέλος του δεύτερου χρόνου και από ό,τι φαίνεται ε, ο στόχος μας θα πετύχει. Αυτό σημαίνει ότι η κεφαλουαχική αυτή αύξηση στην ουσία λειτουργήσε σαν για 200 ε, περίπου ε, δις. Το θέμα είναι βέβαια αν ε, φτάνουν τα ποσά αυτά. Φυσικά και βοηθούν τα ποσά αυτά, όπως είπε και ο Ιρλανδός Ευρωβουλευτής, όταν βρίσκεται κανείς στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται η τράπεζα, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Βέβαια αυτό δεν αρκεί. Αν κάποιος αναρωτηθεί, προφανώς και κάτι τέτοιο δεν είναι επαρκές υπάρχουν ε, ε, κάποια τεράστια κενά τα οποία δεν καλύπτονται. Υπάρχει καταρχάς ένα τεράστιο κενό σε ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες ε, υποδομών επενδυτικού τύπου. Και υπάρχει επίσης Υπάρχει λοιπόν και άλλο ένα κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα τις σχέσεις επένδυσης και καινοτομίας. Έχουμε αρχίσει και μένουμε πίσω τα τελευταία χρόνια στα επενδυτικά μέσα στην καινοτομία. Αυτό σημαίνει επένδυση στην ανταγωνιστικότητα. Έχουμε επίσης και μια πολύ μετριασμένη όρεξη επενδυτική στον ιδιωτικό τομέα οι τράπεζες του ιδιωτικού τομέα αποστρέφονται τον κίνδυνο πλέον. Και γι' αυτό ε, τα περιθώρια τα οποία συνολικά έχουμε είναι περιορισμένα. Αν τα σωρεύσετε όλα αυτά βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα επιτρέψει την μεταφορά της υπάρχουσας στην αγορά ρευστότητα στις πραγματικές επενδύσεις. Και αυτή η πλατφόρμα είναι κάτι που μας απασχολεί. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέποντας τα ιδιωτικά κεφάλαια να αναλάβουν να διατρέξουν περισσότερους κινδύνους έτσι ώστε να διευκολύνουν την οικονομία, τη λειτουργία της οικονομίας. Αυτό μας απασχολεί στην παρούσα και νομίζω ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον επόμενο μήνα θα κάνει ακριβέστερες προτάσεις. Επίσης, Υπάρχουν κάποια επιμέρους σημεία τα οποία έχουν τεθεί από τους συναδέλφους σας στα πλαίσια της ανάλυσης την οποία έχει κάνει μέχρι τώρα ο εισηγητής σας. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλά κάνετε και συγκεντρώνετε την προσοχή σας. Αντιπροσωπεύουν το 80 με 85% της απασχόλησης στην Ευρώπη οι μικρομεσαίες. Ως εκ τούτου αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας και της οικονομικής ανάκαμψης. Εμείς φυσικά αυξήσαμε τις δραστηριότητές μας από 14 δις ε, τον προπροηγούμενο χρόνο πήγαμε στα 22 εφόσον λάβετε υπόψη σας και το IMF. Ε, προφανώς και δεν επαρκούν τα ποσά αυτά υπάρχουν κάπως διαφορετικές εκτιμήσεις, αλλά υπάρχει ε, μια ζήτηση η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερη και 20 φορές μεγαλύτερη λέγουν ορισμένοι από το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πιο αποδοτικοί και στα πλαίσια της εκτέλεσης του προγράμματος Juncker. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε ιδιαίτερα είναι ο τομέας της ενέργειας και της ε, αποδοτικότητας της ενέργειας. Όπως γνωρίζετε και όπως υπόθηκε επανειλημμένα, εμείς έχουμε περίπου το 27% των επενδύσεών μας που ε, οδεύουν σε δραστηριότητες αποδοτικότητας της ενέργειας και αντιμετώπισης των κλιματολογικών συνεπειών και οι επενδύσεις μας εκτός Ευρώπης είναι σε αυτόν τον τομέα περίπου το 30% του συνόλου των εξωτερικών επενδύσεων. Εμείς δεσμευόμεθα φυσικά από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, των εκπομπών καυσαερίων καλύτερα και έχουμε επίσης ε, βάλει και κάποια νέα στάνταρντ ε, επιδόσεων που αφορούν όλα τα προγράμματα ε, με ορυκτά καύσιμα και των οποίων οι εκπομπές ξεπερνούν ένα κάποιο επίπεδο, ένα κάποιο ύψος. Η δράση μας λοιπόν στον, κλιματικό τομέα είναι βασική, ε, βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Όπως επίσης γνωρίζετε ή έχετε παρατηρήσει, εμείς κάναμε και μία δήλωση επίσημη για την δράση μας στον τομέα των περιβαλλοντικό εδώ και ένα χρόνο και έχουμε ξεκινήσει να, και θα ξεκινήσουμε μάλλον να αξιολογούμε εκ νέου τη στάση μας γύρω από τα θέματα αυτά ήδη από το 2015. Θα προηγηθεί μια νέα διαβούλευση η οποία μάλιστα όπου να είναι θα ξεκινήσει. Λοιπόν, σε ό,τι έχει σχέση με την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με πιο ε, ικανοποιητικό τρόπο. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει ένα κύμα ετοιμάτων στα πλαίσια του, του προγράμματος Juncker, ε, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια περισσότερο. Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο θέσατε αρκετοί από σας αφορά την όρεξη σε εισαγωγικά την οποία έχουμε για να αναλάβουμε κινδύνους. Κάποιοι πιστεύουν ότι έχουμε ανοιχτεί αρκετά, άλλοι πιστεύουν το αντίθετο. Να σας εξηγήσω πώς το βλέπουμε εμείς το θέμα αυτό της εκθεσης κινδυνο εκείνη. Εμείς έχουμε ένα επίπεδο 3α. Αυτό δεν είναι φετίχ βέβαια δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να είμαστε μόνον υπερήφανοι, αλλά έχει μια λογική το ότι εμένουμε σε αυτό. Έχοντας αυτό το καθεστώς 3α μπορούμε να δανειστούμε ευθυνότερα στις αγορές ε, και δανειζόμενοι ευθυνά μπορούμε φυσικά να δώσουμε χαμηλά επιτόκια στον καταναλωτή. Αν αυξηθεί το κόστος δανεισμού μας τότε φυσικά κάποιοι από τους καταναλωτές μας, εισαγωγικά καταναλωτές, θα χάσουν κάποια από τα πλεονεκτήματα της, του χαμηλού κόστους ε, το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα. Και σε σχέση με τους επενδυτές, όπως ξέρετε πρέπει να προσφέρουμε στις αγορές σε αιτήσια βάση για να παίρνουμε κάποια χρήματα, 70 με 80 δις σε αιτήσια βάση. Κάποιοι από τους επενδυτές χρειάζονται ένα τμήμα επενδύσεων να ανήκει σε επενδυτικά προϊόντα 3α για να μπορέσουν να δώσουν τα χρήματά τους. Και γι' αυτό αν εμείς κατέβουμε θα είναι πιο δύσκολο να βρούμε τα χρήματα αυτά. Και ξέρετε ότι η μισή περίπου από τους επενδυτές των ομολόγων που εμείς εκδίδουμε δεν είναι Ευρωπαίοι επενδύουν επειδή αγαπούν την Ευρώπη, αλλά βασικά επενδύουν γιατί θέλουν να έχουν μια ασφαλή και παραγωγική επένδυση για τα χρήματά τους. Και μια τελευταία παρατήρηση. Έγιναν αρκετές παρατηρήσεις, τις οποίες εξετίμησα δεόντως για τα ομόλογα έργου, για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται με τα project bonds. Εμείς βρισκόμαστε στο μέσο της πιλωτικής, της προπαρασκευαστικής φάσης. Μόνο πέντε προγράμματα έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα και κάποια άλλα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση και βρίσκονται στις αντίστοιχες φάσεις. Αλλά η πιλωτική αυτή φάση, όπως και το είχαμε πει, εμπλέκει τομείς όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές. Όπως επίσης γνωρίζετε, και αυτό δεν θα εκπλήξει κανέναν από εσά, στα πλαίσια αυτής της πιλωτικής φάσης υπάρχει μια ε, τακτική παρουσίαση της κατάστασης αναεξάμεινο, όχι μόνο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και προς εσάς, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το κάνουμε αυτό έτσι ώστε να σας δείξουμε το σε ποια φάση βρισκόμαστε κάθε στιγμή. Και όπως είπα, αυτή η πρωτοβουλία, το PPI για τα, έργα, τα ομόλογα έργων, υπόκειται σε συγκεκριμένα επίπεδα αν θέλετε αυστηρότητας, προστασίας, εποπτείας και ελέγχου και αξιολόγησης όπως και όλες οι άλλες τράπεζες. Και τίθεται επίσης εδώ ένα επιπλέον θέμα και το θέμα της συμμόρφωσης. Είναι λοιπόν όλα αυτά σε σχέση με τα PPI θέματα τα οποία δεν είναι εκτός διαδικασιών ελέγχου αλλά παραμένουμε υπόλογοι όπως και σε όλα τα άλλα στα πλαίσια των PPI. Όπως ξέρετε έγινε μια εξωτερική ελεγκτική αξιολόγηση για την πιλωτική φάση. Η αξιολόγηση αυτή εξέτασε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί και την έκρινε ικανοποιητική έχει προτείνει επίσης και κάποιες αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα μελλοντικά μέσα τα οποία θα δημιουργήσουμε και όπως επίσης γνωρίζετε ε, ο έλεγχος αυτός είναι πλέον διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα μας. Έχουν υπάρξει λοιπόν ε, κάποιες πιο συγκεκριμένες αναφορές στο πρόγραμμα Κάστορ. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ε, το έχω συζητήσει άλλωστε μεμονωμένα με πολλούς από εσά. Πάντως να έχετε υπόψη σας ότι εμείς ακολουθούμε επακριβέστατα τις ίδιες διαδικασίες τις οποίες ακολουθούμε και με άλλα προγράμματα. Ό,τι κάνουμε δηλαδή στα άλλα προγράμματα το κάνουμε και στα PPI. Κλείνοντας, λέει ο μιλητής για τρίτη φορά, έχουν γίνει ορισμένες παρατηρήσεις για το θέμα της συμμόρφωσης και για το θέμα της διαφάνειας. Να πω ότι έχουμε ένα μηχανισμό ελέγχου συμμόρφωσης ο οποίος θα έλεγα είναι ιδιαίτερος εκτεταμένος. Είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου σε τακτική βάση ε, κάνουμε συναντήσεις συνοδητοποίησης του συγκεκριμένου θέματος όχι μόνο στο εσωτερικό της τράπεζας αλλά και με οργανώσεις εκτός και είναι κάτι το οποίο έχει θα έλεγα συνεισφέρει σταδιακά σε μια καλύτερη συνειδητοποίηση του θέματος σχετικά ε, με την λογοδοσία μας. Είμαστε στο μέσο ε, μιας διαδικασίας αναθεώρησης για μια ακόμη φορά του μηχανισμού παραπώνων, ε, μέσω του μηχανισμού που έχουμε, ξέρετε ότι έχουμε τακτικές ακροάσεις, ήδη η επόμενη θα γίνει το Φεβρουάριο, και συνεργαζόμαστε στενά και με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό γιατί έχει σχέση με τον έλεγχο της τραπεζάς μας και με τον τομέα και για τον τομέα της διαφάνειας είσαστε επίσης εν γνώση ότι έχει προηγηθεί μια διαβούλευση για την αναθεώρηση της πολιτικής μας που ξεκίνησε εδώ και μισό περίπου χρόνο Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να καταστήσουμε την πολιτική μας στον τομέα της διαφάνειας πιο ε, συγκεντρωμένη και πιο αναγνώσιμη ε, και καλύτερα εντασσόμενη στο κοινοτικό πλαίσιο. Ε, εμείς έχουμε συνδεθεί επίσης και με την διεθνή προσπάθεια διαφάνειας. Είμαστε ένας από τους πρώτους διεθνείς οργανισμούς που συνδεθήκαμε μαζί τους και ελέγχονται τα θέματα της διαφάνειας σε χρηματοδοτήσεις που πηγαίνουν σε προγράμματα εκτός των συνόρων της Ένωσης. Λοιπόν, αυτά δεν έχω άλλου είδους γενικές παρατηρήσεις. Αν όμως εσείς έχετε περισσότερες ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, παρακαλώντας τον να είναι σύντομο, διότι δαπανίσαμε πολύ περισσότερο χρόνο για αυτό το θέμα δεν είχαμε την έκτα, αλλά τέλο πάντων το επόμενο σημείο πρέπει να ξεκινήσει ακριβώ στι 5. Όταν σου τότε θα ευχαριστήσω απλά και μόνο όλου ε, όσου ε, προέβησαν σε σχόλια. Πιστεύω ότι Υπάρχει, πιστεύω, κάποια γενική συνένεση επί τη οποία μπορούμε να εργαστούμε. Συμφωνείτε όλοι, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή ε, της ΕΤΕΠ και των μέσων της και πρέπει να διευρυνθούν αυτά για να μειωθεί το κενό των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω συμφωνούμε επίσης ότι η έκθεση δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με όλη τη δεσμευμένη τον Γιούγκερ, αυτό θα πρέπει να γίνει σε μια ξεχωριστή έκθεση, αλλά στο ρόλο τη ΕΤΕΠ να επικεντρωθεί. Σημαντικό είναι και ο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Σνάσο από το ΕΛ και πολλοί άλλοι είπαν ότι θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στι ΜΜΕ. Συμφωνώ και προσβλέπω στι προτάσει σα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους αφορολογικού παραδείσους που έθεσε ε, από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, ναι, νομίζω ότι μπορούμε να ε, αναφέρουμε κάποια πράγματα στην ε, έκθεση και νομίζω ότι και η κοινή γνώμη θα είναι στο πλευρό μας. Τώρα το θέμα της λογοδοσίας, πράγματι αναφέρονται τα σχετικά και η τοπική κοινωνία, η τοπική φορείς όπως είπε η Στάσο και η συμμετοχή τους θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη. Είναι μια σημαντική τροπολογία. Συμφωνώ και σε ό,τι αφορά τα ομόλογα έργων πολύ τα αναφέρατε συνάδελφοι από την ΚΟΥ, από την ε, EFTD, με τα ομόλογα εργών ε, ξέρουμε ότι είναι σε αυτή την πιλωτική φάση. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει μια κριτική αξιολόγηση του μηχανισμού. Θέλουμε και η τράπεζα να μελετήσει το μηχανισμό αυτό, γιατί κάποιες φορές ε, υπήρξαν ενστάσεις με ορισμένα μεγάλα έργα σε κάποιες χώρες. Καλό είναι λοιπόν να ζητήσει το Κοινοβούλιο από την τράπεζα να τα εξετάσει όλα αυτά γιατί αναφέρεται μόνο το έργο Κάστο. Ε, απλά γιατί είναι το πρώτο, γι' αυτό αναφέρεται στην έκθεση, δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο. Μπορούμε να το συζητήσουμε πάντω έτσι περαιτέρω. Μου άρεσε πολύ επίση το έτοιμο ε, να ληφθεί υπόψη το ότι μόνο μία είναι η γυναίκα μέλος ε, του Διοικητικού του Συμβουλίου Διοικητών. Δεν με ακούει τώρα δυστυχώς η κυρία που το ανέφερε, αλλά ε, είναι πολύ καλή ιδέα της και επειδή τελειώνει ο χρόνος, Θέλω να πω απλά στον εκπρόσωπο της ΕΤΕΠ εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ παρόντι σήμερα. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας ε, και ευχαριστούμε την τράπεζα για την υποδοχή στο Λουξεμβούργο. Η μερίδα εργασίας εκεί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική. Θέλω τέλος να πω ότι στην αξιολόγησή μας προσπαθούμε να εκφράσουμε ε, τις θετικές μας εκτιμήσεις απέναντι στα θετικά βήματα που έχει κάνει η τράπεζα. Επίσης πολλές φορές λέμε ότι καλωσορίζουμε, χαιρετίζουμε διάφορες δράσεις για τη λογοδοσία κτλ. Και ο ρόλος του Κοινοβουλίου όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι να ασκεί κριτική. Να βλέπουμε κριτικό μάτι τα σχετικά. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρούμε χρόνο να κάνουμε μια πιο διεξοδική σε βάθος συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το χρονοδιάγραμμα 15 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, θα εξετάσουμε τις τροπολογίες 8 Ιανουαρίου, 27 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και τέλος Μαρτίου προβλέπετε στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Να χαιρετήσω τώρα τον ε, υποψήφιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε, ώστε να ξεκινήσουμε την δημόσια ακρόαση της υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης. Χαιρετίζουμε την Δόκτορα Έλκε Κιόνιχ. Είναι η πρόεδρος της ε, Ομοσπονδιακής Αρχής Εποπτείας στην Γερμανία, η Δόκτωρ Κιόνικ έχει επιλεγεί από την Κομισιόν <clears throat> ως υποψήφια για τη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Εξυγένσης, του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγένσης μάλλον. Είχαμε ήδη την ευκαιρία να έχουμε μια κεκλεισμένο των θυρών ε, στις 16 Νοεμβρίου μια συνάντηση με την κυρία Κιόνικ από τη στιγμή που ήταν ήδη στον περιορισμένο κατάλογο υποψηφίων από την Κομισιόν. Την ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία της και στο άτυπο στάδιο της διαδικασίας που έδωσε δυνατότητα στους, στα μέλη της Επιτροπής να αξιολογήσουν τους υποψηφίους και την ευχαριστούμε που είναι και τώρα ενώπιόν μας στη δημόσια αυτή ακρόαση η οποία παίζει ένα σημαντικό ρόλο για να υπογραμμίσει τον χαρακτήρα λογοδοσίας του Ταμείου του Συμβουλίου Εξυγίανσης και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα μέλη της Επιτροπής μας. Όπως τα γνωρίζετε, η Επιτροπή μας θα συναντηθεί και αύριο το πρωί σε έκτακτη συνεδρίαση για, αλλά και αυτή θα είναι ε, δημόσια και θα μεταδίδεται στο διαδίκτυο για να ακούσουμε τους πέντε υποψηφίους για την Αντιπροεδρία και τις άλλες θέσεις του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγένσης. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη δημιουργία αυτού του νέου εργαλείου της Τραπεζικής Ένωσης και σημαντικά για την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο το οποίο έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στην δημιουργία αυτού του μηχανισμού ενίας εξυγίανσης και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εκπρόσωποι του Ευρωπαίου πολίτες, πολίτη έπαιξε σημαντικό ρόλο στο διορισμό των μελών και του Προέδρου του Συμβουλίου Εξήγησης. Δίνω το λόγο λοιπόν στην κυρία Κιόνιγκ για 7 λεπτά για την εισαγωγική της παρέμβαση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη, <clears throat> νιώθω μεγάλη τιμή και είναι πραγματικά ένα προνόμιο για μένα να μπορέσουν να έλθουν ο σας και πάλι για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγένσης και για το σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να αναλάβει στο μέλλον. Το, ο μηχανισμός εξυγένσης είναι ο λογικός δεύτερος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης, όπως και ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο μηχανισμός εξυγίανσης που βασίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών θα πρέπει να αλλάξει την κατάσταση στο τραπεζικό τομέα και θέλω ιδιαίτερα να συμβάλλω σε αυτό. Όταν συστημικά σημαντικέ τράπεζε αντιμετωπίζουν δυσκολίε, στο μέλλον θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην εξυγίανσή του με έναν τρόπο ο οποίο είναι τακτικό. Χωρί κίνδυνο προς την κοινωνία ως σύνολο και χωρίς να χρειαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη ο φορολογούμενος. Και έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα άλλα μέσα τα οποία ευτυχώ είναι στη διάθεσή μας. Θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία του bail-in, της συμμετοχής δηλαδή των ομολογιούχων και όχι το bail-out, η χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα. Το ε, Συμβούλιο Εξυγείας θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτό γίνεται σωστά και με την σωστή κατανομή στο βάρους. Αυτή είναι μια πρόκληση που είμαι έτοιμη να αναλάβω. Με το σύστημα αυτό ελπίζουμε θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα τα οποία είναι αλληλένετα. Καταρχήν δεν θέλουμε μια άλλη περίπτωση Lehman Brothers. Θέλουμε να απελευθερωθούμε από την υποχρέωση πραγματική υποτιθέμενη του να αποφύγουμε αντίστοιχε περιπτώσεις όπως ήταν αυτή των Lehman Brothers με το να διατηρούμε εν ζωή τράπεζες με λεφτά φορολογουμένων. Τονίζουμε λοιπόν μια βασική αρχή της οικονομίας της αγοράς η οποία είχε τα ανασταλεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι οι τράπεζες όπως και οι άλλες επιχειρήσεις έχουν ευθύνη για τις ενέργειές τους. Και εδώ είναι το μεγαλύτερο πλέον έκτημα της ε, οδηγίας για την ε, ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών και του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης. Ο στόχος δεν είναι λοιπόν να κάνουμε μια χιδία πολυτελή για τα μεγάλα συστημικά σημαντικά πιστοτικά ιδρύματα. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα με το να εφαρμόζουμε με προδραστικό τρόπο τη δυνατότητα εξυγίανσης των τραπεζών. Με έναν τρόπο ο οποίος είναι αξιόπιστος και επομένως έχει και ένα αποτρεπτικό χαρακτήρα και μπορεί να εξασφαλίσει την πειθαρχία των πιστοτικών ιδρυμάτων. Θα πρέπει να γίνει σαφές προς τις τράπεζες και προς τους πιστωτές τους ότι δεν μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξη του ε, την κρατική υποστήριξη εάν αποτύχει το μοντέλο, επιχειρηματικό της μοντέλο. Η σωστή σχεδίαση της εξυγένσης εξασφαλίζει ότι το Συμβούλιο Εξυγένσης θα μπορέσει να συμβάλλει στην εξυγένση εγκαίρως. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρξει μια ομαλή αλληλεπίδραση μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης, των Εθνικών Αρχών Εξυγίανσης, του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου ο σχεδιασμός της εξυγένσης θα πρέπει να είναι αναλογικού χαρακτήρα, να λάβει υπόψη το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των ιδρυμάτων που πρέπει να εξηγιαθούν. Αν όμως ένα τέτοιο πιστοτικό ίδρυμα είναι σε κατάσταση αστοχίας, είναι πιθανή η αστοχία του, θα πρέπει να εξασφαλίσει ο μηχανισμός αυτός την ισότητα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση μεταξύ χωρών και τραπεζών. Και αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από το Ταμείο Εξυγίανσης, θα πρέπει να το πράξουμε. Αλλά δεν θα πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να φτάσουν μέχρι αυτού του σημείου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι τράπεζε διατηρούν σημαντικά και επαρκή ίδια κεφάλαια, ώστε τα κεφάλαια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εξυγίανση και οι απώλειες θα πρέπει να τι επομιστούν οι ομολογιούχοι και οι μέτοχοι και θα πρέπει να γίνει η μεταρρύθμιση και η αναδιάθρωση της τράπεζας ώστε να μπορεί να υπάρχει εξυγίανσή της με ομαλό τρόπο. Δεν πρόκειται λοιπόν για ανάνυψη των τραπεζών αλλά για αναδιάθρωσή τους. Και εδώ υπάρχει στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση η υποχρέωση για ένα ε, ελάχιστο επίπεδο ιδίων ε, κεφαλαίων MRL όπως λέγεται στα αγγλικά. Με την πρότασή της για τη συνολική ικανότητα απορρόφησης απολειών, TILAC την αργό, το Συμβούλιο ε, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά προχωρεί και ένα βήμα παραπάνω. Επιπλέον, θα χρειαστούμε κανόνες για να εξασφαλίσουμε την παροχή ρευστότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγένσης, ώστε να μην χρειαστούμε <clears throat> να υπάρξει από το δημόσιο κορβανά υποστήριξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει και το Ταμείο ε, σταθερότητος και επίσης έχει ξεκινήσει να γίνεται και σε επίπεδο του, ε, ενία, του Συμβουλίου Ενίας Εξήγενσης. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα τα οποία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά με ένα συνολικό σύστημα εξήγενσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δράξουμε ως ένα σημαντικός ευρωπαϊκός εταίρος διαπραγμάτευσης και να συμβάλλει στο να υπάρξει ένα συνολικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σύστημα εξυγίανση και οι αρμόδιες πρακτικές. Είμαι έτοιμη να προχωρήσω πως αυτή την κατεύθυνση μαζί με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου ε, Εξυγίανση και με όλους τους άλλου εμπλεκομένου. Και αυτό περιλαμβάνει την καλή συνεργασία μεταξύ των, ε, της μητρικής εταιρείας και των ε, τοπικών αρχών για να γίνει σωστά αυτή η διαδικασία εξυγίανσης. Και το πιο σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των τραπεζών και των αρχών. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ, αφού τονίσω και πάλι ότι εσείς ως μέλη του Κοινοβουλίου, ως εκπροσωποί εκλεγμένοι των Ευρωπαίων πολιτών, θα παρακολουθήσετε από πολύ κοντά το έργο του Μηχανισμού Εξυγένσης και του Συμβουλίου, του Ενίου Συμβουλίου Εξυγένσης. Είμαστε υπόλογοι σε εσά και αυτό κατά την άποψή μου είναι απαραίτητο και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ δόκτωρα Κένι. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τα λόγια σας για την ε, λογοδοσία του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βασιζόμαστε σε αυτό. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρώτο μιλητή, τον κύριο Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είσαστε πάλι μαζί μας ενώπιον της Επιτροπής μας. Δύο ερωτήματα έχω να σας θέσω. Καταρχήν, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάτι που το έχω αποκομίσει και από τη δική μου εμπειρία στην εκλογική μου περιφέρεια και από άλλες εκλογικές περιφέρειες όπου έχω βρεθεί. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται τώρα με την εξυγίανση τραπεζών. Οι φορολογούμενοι θα χρειαστεί και πάλι να πληρώσουν για κάποια εξυγίανση τράπεζας ή για μια διάλυση τράπεζας, για μια εκαθάριση. Και επίσης θα υπάρξει κάποια αρχή μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα είναι αρμόδια για αυτήν την διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό για τη δική σας ανεξαρτησία εναντί της Ευρωπαϊκής Κομισιόν και πώς θα αποχωριστεί η δική σας αρμοδιότητα από αυτήν της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Κιόνιχ. Θα σας απαντήσω φυσικά στα γερμανικά. Το πρώτο ερώτημα είναι κατά πόσο θα συντηθεί και πάλι από τους φορολογούμενους να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αν θα είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είμαστε σωστοί στο σημείο αυτό. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Έχουμε τράπεζες οι οποίες είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες. Έχουμε το μηχανισμό εποπτείας για τις μεγάλες τράπεζες, τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, τον οποίο δημιουργούμε. Αλλά εγώ θα πρέπει να ήμουν, θέλω να είμαι πολύ επιφυλακτική. Δεν μπορώ να σας πω ποτέ πια δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο δεν θα υπάρχει ανάγκη για χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους. Ελπίζουμε ότι έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο και ότι θα έχουμε πολλά επίπεδα άμυνας προτού φτάσουμε και πάλι στο φορολογούμενο. Δεν σας πω, δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Μπορώ να σας πω όμως ότι είμαστε καλύτερα οργανωμένοι και καλύτερα εξοπλισμένοι. Έχουμε κάνει πολλές κινήσεις προς την, την καλή, τη σωστή κατεύθυνση ώστε να γίνει πολύ πιο απίθανη προσφυγή στους φορολογούμενους ανεξαρτησία από την Κομισιόν ή γενικά η ανεξαρτησία του από το μηχανισμό εποπτείας. Η δική μου εμπειρία <clears throat> είναι ότι η καλύτερη λύση εδώ είναι να είμαστε ανεξάρτητοι με το να πούμε ποια είναι η δική μας θέση ως ε, οργανισμός να ακολουθούμε μια σαφή γραμμή και να προσπαθούμε να πείσουμε και τους άλλους με επιχειρήματα τα οποία είναι γνωστά. Εσείς γνωρίζετε τη γερμανική πραγματικότητα όπου είναι το Γερμανικό Υπουργείο ε, Οικονομικών αυτό το οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Εγώ έχω εργαστεί εκεί ανεξάρτητη ως πρόεδρος της BaFin, της Εποπτικής Αρχής για τα Γερμανικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και έχω κάθε ελπίδα ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η παράδοση. Σε ευχαριστώ για την ομάδα των Σοσιαλιστών ο Φων Βαϊσέκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κένιχ, διαρωτώ με. Μετά από τον προλαλήσαντα συνάδελφο. 55 δις είναι το, το ταμείο. Αρκεί αν έχουμε ε, έντονες πιέσεις αν δείτε και τη βιβλιογραφία με τις τραπεζικές κρίσεις, λέτε ότι θα έχουμε και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Μιλάμε ίσως για ένα 20% του ε, ΑΕΠΑ που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι 20 40 φορές περισσότερο από το Ταμείο των 55 δις που καλύπτει μια οκταετία. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι στην πραγματική ζωή αυτά τα στοιχεία είναι λογικά αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον μια σοβαρή συστημική τραπεζική κρίση. Και με βάση το αξίωμα για το οποίο θα τους επεθοριστείτε. Απάντηση. Καταρχάς, η απάντηση η πρώτη που έχω να δώσω είναι ότι πρέπει στο σχεδιασμό μας ό,τι αφορά την εξυγίανση ε, να προκαταλαμβάνουμε τις εξελίξεις και όχι να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αμέσως. Πώς γίνεται αυτό, να έχουμε πιο ασφαλές τράπεζες. Και το Σαββατοκύριακο χαμογελούσα γιατί έλεγε ότι αν ο ενιαίος εποπτικός ε, μηχανισμός λειτουργήσει το Συμβούλιο Εξυγίανσης ε, θα είναι πολύ μοναχικό. Τέλο πάντων, αστείευομαι. Σίγουρα θα έχουμε πολύ στενή συνεργασία και από πολύ νωρί θα συμμετέχουμε στη διαδικασία για να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε ένα επικείμενο πρόβλημα. Βέβαια, πάντοτε μπορεί κανείς ε, να κάνει υποθέσει για το ύψος του κεφαλαίου που μπορεί να χρειάζονται οι τράπεζες. Κάποιοι ακαδημαϊκοί ζητούν το 30%. Ε, και πρέπει να σας πω ότι ε, στα τέλη του 10ου αιώνα είχαμε κρίση παρότι υπήρχε αυτό το κεφάλαιο τότε στράψη 30% δεν είναι το κεφάλαιο το μόνο επιχείρημα, το ίδιο ισχύει και για το ταμείο. Λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι το ταμείο αυτό ε, θα τροφοδοτηθεί με αυτά τα ποσά από την επόμενη οκταετία, εγώ πιστεύω ότι η ιδέα είναι καλά θα μπορούσαμε να δούμε και το ενδεχόμενο δανειοληψίας. Κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται να το αγγίξει κανείς αυτό, αν έχει κάνει σωστά το σχεδιασμό εξυγίανσης. Αν τώρα ε, γκρεμιστούν όλοι οι φούρνοι και πεθάνουν όλοι οι λύκοι, ε, μπορεί να συμβεί. Ε, αυτό που λέτε να ήταν μια καλή λύση. Thank σε ευχαριστώ πολύ. Λούκε. Uh, Κυρία Κιονίχ, καλώς ήλθατε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι εσείς έχετε δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσετε την, ε, τη συμβολή των ε, ε, φορολογουμένων ή να την μηδενίσετε παρά το γεγονός ότι Συμμερίζομαι το σκεπτικισμό του κυρίου Φοντ Βάισέκερ, αλλά αν ακολουθήσουμε την οδό του bail-in, ξέρουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση μπορεί και πάλι να υπάρξει αρνητική επίπτωση για τους ε, φορολογουμένους, παραδείγματος χάρη μέσω των συνταξιοδοτικών ταμείων ή των ασφαλιών, όπου ουσιαστικά η, αποταμίευση των ε, πολιτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασώσει μεγάλες τράπεζες. Το ερώτημα προς εσάς τώρα είναι το εξής. Όταν μιλάτε για την ανάγκη να έχουμε προδραστικές λύσεις, φανταζούμε ότι αυτό σημαίνει ότι είσαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε και τους μηχανισμούς του bail-in. Να δείτε λοιπόν για κάθε τράπεζα σε ποιο βαθμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός σε περιπτώσεις κρίσης. Εσείς θέλετε τώρα να πληροφορήσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δική μας Επιτροπή σε ποιο βαθμό θα υπάρξει και η υποχρέωση και για επενδυτές οι οποίοι είναι πολιτικά ευαίσθητοι μέσα σε εισαγωγικά και θα τους ζητηθεί η συμβολή τους και πώς, εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κληθούν κάποιοι άλλοι να αναλάβουν την ευθύνη της υποστήριξης. Δηλαδή, αν μπορείτε να μας πείτε ποιο θα είναι το ποσοστό που θα πρέπει να ζητηθεί από τέτοιους ευαίσθητους φορείς στην περίπτωση ανάγκης διάσωσης μιας τράπεζας. Μέχρι ποιου σημείου θα πρέπει να συνεισφέρουν. Εγώ σας δίνω δίκιο γιατί όταν λέτε ότι για τα στοιχεία του Μπέιλιν θα πρέπει να σκεφτούμε τρία πράγματα. Τι πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε τράπεζα. Δεύτερον, ποια είναι η ποιότητα αυτού του κεφαλαίου. Δεν είναι μονάχα ο όγκος, αλλά και το είδος του κεφαλαίου που θα είναι διαθέσιμο και επίσης το ερώτημα ποιος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του αυτά τα στοιχεία. Φυσικά, σε όλες τις διαδικασίες στο τελικό στάδιο υπάρχει πάντα ένας καταναλωτής. Στο τέλος της αλυσίδας υπάρχει πάντα ένας ε, καταναλωτής, ένας φορολογούμενος. Γι' αυτό τονίζουμε την ανάγκη να υπάρχει ένα μεγάλο ύψος στα ταμεία αυτά. Θέλουμε να έχουμε την ποιότητα αυτών των ε, κεφαλαίων και επίσης να έχουμε και κάποιους ε, προσδιορισμούς για το ποιοι φορείς θα πρέπει να έχουν αυτά τα στοιχεία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό με ένα τέτοιο τρόπο που να κινδυνεύουμε να ξεκινήσουμε μια αλυσιδωτή αντίδραση και επομένως δεν προχωρούμε στην εξηγένση γιατί φοβόμαστε τι θα γίνει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά θα πρέπει να συμβάλλει στην ε, σκέψη του ποιοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται και ποια ιδρύματα θα πρέπει να συμβάλλουν στο να κρατούν το κεφάλαιο αυτό που είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ κυρία Κένιχ. Χαίρομαι πάρα πολύ που εν, μέρη έχετε διαψεύσει την ε, καγκελάριο της Γερμανίας η οποία είπε ότι ποτέ πια δεν θα χρειαστεί ο φορολογούμενος να συμβάλλει. Στο σημείο αυτό ήσασταν πολύ πιο πιστικοί. Θέλω να αναφερθώ σε ένα σημείο τώρα σε αυτά που είπατε. Συζητάτε στην Ευρώπη το θέμα της, ε, του χωρισμού των δραστηριοτήτων των τραπεζών μέσα στην διαδικασία αλλαγής των κανόνων για τις ε, τράπεζες και φαίνεται να έχει μειωθεί η ζέση της Κομισιόν να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρείτε εσείς ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σωστό να γίνει μια τέτοια διαδικασία ε, διαχωρισμού των δραστηριοτήτων των τραπεζών και είναι απαραίτητο για τη φιλοδοξία της Κομισιόν. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε την συζήτηση για τις τράπεζες σε σχέση με τα λεγόμενα cash commitments, δηλαδή να υπάρχει μια δέσμευση για την καταβολή ε, ε, χρημάτων από τις τράπεζες και να θεωρείτε ότι δεν είναι μόνο οι τράπεζες υποχρεωμένες να καταβάλουν αυτά τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Υπήρξε αυτή η συζήτηση στη Γαλλία. Για τις ε, αλλαγές, εγώ θεωρώ δεδομένο πάντα ότι αυτοί οι κανόνες, λέει η κυρία Κιόνικ, είναι απαραίτητοι στα πλαίσια της εξασφάλισης της εξυγίαν, του εξυγιαντού των τραπεζών. Να μπορεί δηλαδή μια τράπεζα να περάσει σε μια διαδικασία εξυγίανσης και αυτά περιλαμβάνονται και στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες δομές οι οποίες επιτρέπουν να, να, να γίνεται δυνατή η εξυγίανση. Το θέμα τώρα το οποίο είναι πιο πολιτικό είναι το αν θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των συναλλαγών της τράπεζας για δικό της λογαριασμό με αυτές για λογαριασμό των, των πελατών της. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε μια τέτοια ρύθμιση η οποία ε, έκανε υποχρεωτική να υπάρχουν πάρα πολλές ε, λεπτομερείς ρυθμίσεις. Σίγουρα όμως είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς κανόνες για όλα αυτά. Στους γερμανικούς κανόνες είναι απαραίτητο να μπορούν οι εποπτικές αρχές να επιβάλλουν διαφορετικές αλλαγές στις τράπεζες και όπως έχει λειτουργήσει η δική μας πρακτική, πάντα η αρμόδια εποπτική αρχή μπορεί να το επιτύχει αυτό στις, ε, ε, στη Γερμανία. Τώρα για τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να με τα οποία πρέπει να συμβάλλουν οι τράπεζες στο Ταμείο Εξυγίανσης, Ξέρουμε ότι συνεχίζεται η συζήτηση για τα θέματα αυτά, για το πώς θα πρέπει να συμβάλλουν. Μας ενδιαφέρει να δούμε με ποιο τρόπο αυτά τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα. Αλλά δεν είμαστε ακόμα στο τελευταίο στάδιο αυτής της συζήτησης για να ξέρουμε με, ποια, με ποιο ρυθμό και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να διαθέσουμε αυτά τα χρήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ουρτασούν από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομος θα είμαι. Κάποιες τράπεζες στην Ευρωζώνη από ό,τι δείχνουν τουλάχιστον το κόστος το υψηλό των ομολόγων τους έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα και κινδυνεύουν. Θα χρησιμοποιήσετε εσείς τα μέσα σας έτσι ώστε να καταστήσετε όλες τις τράπεζες να έχουν ικανή ρευστότητα. Θα σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα είναι η βασική προσπάθεια την οποία καλούμε να κάνω. Ε, να έχουμε κάποια προγράμματα εξυγίανσης τέτοια τα οποία θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες και των μεγάλων τραπεζών, τις λεγόμενες too big to fail. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε όλες τις χώρες και μερικές φορές θα μας απασχολήσουν τέτοια φαινόμενα και εκτός Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. βάλει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση σύντομα. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια τεράστια έκθεση για τις μεγάλες ε, γερμανικές τράπεζες που φτάνουν τα 3-3 ε, και το το ευρωπαϊκό είναι το γερμανικό μάλλον α, για μια στιγμή υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα μετάφρασης Λοιπόν, ξανά θα πρέπει να ξαναθέσει την ερώτηση του ομιλητή. Στον προϋπολογισμό του 2013, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες ε, φαίνεται ότι έχει ε, μία τεράστια έκθεση σε παραγόγα στην ουσία ξεπερνάει ε, το ΑΕΠ του συνολικά της Ευρώπης. Ε, μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από αυτά τα μέσα. I we never, Κοιτάξτε, εμείς δεν συζητάμε μεμονωμένα την κάθε τράπεζα, αλλά όπως είδα, είπα και στον κύριο Μπάλτς, προσπαθούμε να πάρουμε τα μέτρα έτσι ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι όταν υπάρχουν μεγάλες τέτοιες τράπεζες οι οποίες αντιμετωπίζουν κινδύνους. Εμείς προσπαθούμε με σταδιακό τρόπο να καταστήσουμε όλα τα πιστοτικά ιδρύματα ασφαλέστερα και αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο τις διαφορετικές περιπτώσεις έλλειψης ρευστότητας που μπορεί να υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε λεπτά είναι ο χρόνος για κάθε ερωταπάντηση, εκτός ε, αν έχετε δυνατότητα για το πρόβλημα για δευτερολογία. Ο κύριος Μπερνά Μονό είναι επόμενος. Ε, κυρία υποψήφια, ως πρόεδρος ε, του ενιαίου Συμβουλίου Εξήγησης ε, θα έχετε τεράστια ευθύνη για να επιλύσετε τις ε, συστημικές τραπεζικές κρίσεις που είναι ανεπόφευκτες στην Ευρώπη. Θα πρέπει με το ενιαίο ε, σύστημα εξυγίανσης επίση να ασχοληθείτε. Ποια είναι η αρχή ουσιαστικά, άκρος φιλελεύθερη του Μπέιλιν, δηλαδή οι τράπεζες θα μπορούν ουσιαστικά να δεσμεύουν τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιωτών αποταμιευτών. Ε, ενώ είναι και αυτοί φορολογούμενοι ουσιαστικά. Πρόκειται λοιπόν για μια θεσμική καταστολή αντί να κάνετε την, ε, ε, μια άλλη, αντί να ακολουθήσετε μια άλλη πολιτική της κρατικοποίησης. υπάρχουν διάφορες προτάσεις για το ποσό 100 δις κτλ. Όταν θα είναι επιχειρησιακό μέχρι το 2025 όμως αυτό το σύστημα με τα 55 δις δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο που θα είχαν ε, μαζικές συστημικές κρίσεις, άρα είναι ε, μη επαρκές. Τεχνικό το πρώτο με ρωτήμα, με βάση ποιους κανόνες και από ποιον ε, θα αναλαμβάνετε τη διαχείριση μιας, της κρίσης μιας μη συστημικής τράπεζας εκτός των 130 δηλαδή. Και ποιος θα είναι το δικό σας, ε, το Συμβούλιο ή οι Εθνικές Αρχές θα το διαχειρίζετε αυτές τις περιπτώσεις. Δεύτερον, πώς αντιλαμβάνεστε τη θέση σας. Δηλαδή, εκεί θα είστε για να σώσετε τις ιδιωτικές τράπεζες για να μην μεταδοθεί η κρίση και υπάρξει πιστοτική ασφυξία ή για να προστατεύσετε τους αποταμιευτές για να μην χάσουν ε, τις, ε, τα περισσότερα του στοιχεία όπως συνέβη χθε στην Κύπρο που είχαμε πραγματική ευθανασία των αποταμιευτών. Thank you. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για τις πιο μικρές τράπεζες το ερώτημά σας. Οι εθνικέ αρχέ εξηγήνε θα αναλάβουν ε, τι κρίσει μικρών τραπεζών σε στενή συνεργασία και θα έλεγα και υπό την αιγίδα του ενιαίου Συμβουλίου και μηχανισμού εξυγίανσης. Διπλός είναι ο δικός μας στόχος κατά την άποψή μου. Ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, ίδια πρότυπα σε όλη την Ευρώπη. Αλλά για τις ε, όχι τόσο σημαντικές συστημικά τράπεζες, εκεί οι εθνικές αρχές εξυγένσεις θα αναλαμβάνουν. Το ερώτημά σας διάσωση τραπεζών. Όχι βέβαια, όπως είπα, όποιος εργάζεται σε ένα περιβάλλον πρέπει να φέρει και τον κίνδυνο, το ρίσκο. Δεν είναι ιδιωτικά τα κέρδη, αλλά για τις απώλειες ε, την πληρώνουν οι φορολογούμενοι, ε, πληρώνουν το λογαριασμό. Εμείς θέλουμε και για τους αποταμιευτές, αλλά και για όλο το σύστημα, να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία. Πάντα πρέπει να είμαστε, πιστεύω, προβλεπτικοί και διορατικοί. Καλύτερα να αποφύγουμε την κρίση παρά να έχουμε ένα πλωστάσιο όσο και καλό και αν είναι για να διορθώνουμε εκ των υστέρων την κατάσταση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η Ντανούτα Χούμπνερ είναι η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε όλοι εδώ, πιστεύω και πιστεύουμε ότι δημιουργήσαμε αυτό το μηχανισμό, τον ενιαίο μηχανισμό εξηγήσης, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τέτοια προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά, υπάρχουν πολλοί τομείς ακόμη που είναι πολύ σημαντικοί για την αποτελεσματικότητα γενικά του ενιαίου ε, μηχανισμού εξήγηση και του Συμβουλίου. Όταν δεν υπάρχει αναρμόνιση, δεσπόζουν οι εθνικές ιδιαιτερότητες και από την προηγούμενη θέση σας γνωρίζετε ότι υπήρχαν ε, ευρύτατες, ένα ευρύ φάσμα εποπτικών πρακτικών στην Ευρώπη. Διαφορετικά λογιστικά πρότυπα υπάρχουν και διαφορετικοί συνδυασμοί εποπτικών κανόνων, κρίσεων, ε, οι νόμοι εθνικοί για την αφαιρεγκαιότητα δεν είναι εναρμονισμένοι και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο και τη δουλειά του ενιαίου ε, Συμβουλίου, Συμβουλίου και εθνικέ Αρχές πολλέ φορές είναι διάσπαρτες, μπορεί να είναι ανεξάρτητε, μπορεί όχι και εξού και το ερώτημά μου, σε ποιο βαθμό όλα αυτά τα ζητήματα, εθνικέ ιδιαιτερότητε που υπάρχουν και όλα αυτά, σε ποιο βαθμό μπορεί να παρακολύσουν το έργο σας, να θέσουν προσκόμματα στην καθημερινή λειτουργία του Συμβουλίου και να καταστήσουν το έργο σας αναποτελεσματικό. Αν κληθείτε να κάνετε μια επιλογή, να, να πάρα πολύ γρήγορα κάποιους τομείς που είναι σημαντικοί για τη δουλειά σας, ποιους τομείς θα επιλέγατε. Τους εθνικούς κανόνες περί ή το ενιαίο σχέδιο εγγύης καταθέσεων. Τι θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό στο πλαίσιο της ομοθετικής προσπάθειας για εναρμόνιση, ώστε να μπορείτε να δουλεύετε πιο, με μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία. Απάντηση. Θα ξεκινούσα καταρχάς λέγοντας ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πράγματι διαφορετικές εθνικές πρακτικές ε, στον τομέα της εποπτείας και σε ό,τι αφορά την εξυγίανση, για να μην πω ακόμη πιο πολύ ε, στον τομέα της εξυγίανσης, γιατί πολύ μόλις ξεκινάμε. Και βέβαια όταν μιλάμε για εξυγίανση, οτιδήποτε έχει να κάνει με διαφορετικές ε, ε πρακτικές ε, στον τομέα της αξιολόγησης, εταιρικό δίκαιο ή ε, κανόνες για την αφαιρεγγιότητα. Σίγουρα είναι διαφορετικά, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξη. Βλέποντας και από τον ενό υποπτικό μηχανισμό, ένας χρόνος πέρασε έχουμε ξεκινήσει να συνεργαζόμαστε, μπορεί να μην συμφωνούμε πάντοτε, αλλά κοινό είναι ο στόχος μας και βλέπουμε σε αυτό το χρόνο ότι έχουμε πετύχει πολλά. Ήδη υπάρχει μεγάλη ομοιογένεια. Σίγουρα μακρύ είναι ο δρόμος και για τον ε, νέο μηχανισμό εξυγίανση θεωρώ ότι και εδώ θα πρέπει το δίκτυο των Εθνικών Αρχών εξυγίανση με τη γνώση τους να το αξιοποιήσουμε και να συνδυάσουμε αυτή την εμπειρία με την ευρωπαϊκή προοπτική. Και αυτό θα μας οδηγήσει προς τα εμπρός. Θα ήμουν διστακτική για να σας πω επιλέγω το εταιρικό δίκαιο ή το, τους νόμους για την αφαιρεγγιότητα. Το τελευταίο που είπατε για τις εγγύσεις των καταθέσεων μάλλον δεν θα το διάλεγα. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ένα βασικό μειόμορφο σύστημα που μετά για τις εγγυήσεις ε, των καταθέσεων μπορεί να έχει εθνικές ε, διακλαδώσεις. Το θέμα είναι ότι ήδη έχουμε να κάνουμε πολλά με την οδική για την ανάκαψη και την εξήγηση των τραπεζών. Λύνει διασυνοριακά ζητήματα. Το θέμα είναι τι γίνεται εντό συνόρων και τι γίνεται με τις συστημικές τράπεζες που έχουν κόμπους και στην Ασία και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη. Άρα υπάρχει το διασυνοριακό στοιχείο και εκεί πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Και αυτό μπορεί να γίνει με συμβατικό και όχι τόσο με καταστατικό τρόπο. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ κύριε Σαμπεσάντ. Θέλω να θέσω το ερώτημα του κυρίου Μπαγιέ. Κυρία Κένιχ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας πρότεινε να αναλάβετε την ευθύνη αυτού του οργανισμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ε, των ε, πιστοτικών ιδρυμάτων τα οποία ε, καλείστε να βοηθήσετε. Θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας 55 δις μέχρι το 2024, κατάλαβα καλά. Ο στόχος σας είναι να αποφύγετε νέες χρηματοπιστωτικές κρίσεις στην Ευρώπη. Παρά όμως την ύπαρξη πιο αυστηρών διατάξεων, οι τράπεζες συνεχίζουν να επενδύουν σε τοξικά προϊόντα. Τα στέστρες της Κεντρικής Τράπεζας απέδειξαν τον έφραστο χαρακτήρα των τραπεζών μας. Δύο στις έξι έχουν ακολουθήσει τέτοιου είδους κατευθύνσεις ποια είναι τα συμπεράσματα και τι μπορείτε αντικειμενικά να κάνετε για να φέρετε εις πέρα στην εντολή σας. Αυτή είναι η ερώτηση του κυρίου Μπαγιέ. Πιστεύω πρώτα απ' όλα η δική μου ανάγνωση των ευρωπαϊκών δοκιμασιών αντοχής, stress test, είναι κάπως διαφορετική. Εμείς έχουμε βγει από μια χρηματοπιστωτική κρίση και έχουμε ήδη καταφέρει να προχωρήσουμε. Σύμφωνα ότι υπήρξαν κάποιες τράπεζες οι οποίες απέτυχαν στις δοκιμασίες και τώρα είναι υπό αποκατάσταση, ας το πω έτσι. Αυτό το οποίο είναι η μόνη απάντηση που μπορώ να δώσω, η μόνη λύση που μπορώ να σας προσφέρω, είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του, συμβου, του μηχανισμού εξυγίανσης και του μηχανισμού εποπτείας γιατί η εποπτεία των τραπεζών φυσικά εναπόκειται στον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Και η καλή εποπτεία των τραπεζών αφορά όχι μόνο το κεφάλαιο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των τραπεζών και η αντιμετώπιση των ασθενών τους σημείων. Και η, η σχεδίασή τους λοιπόν μαζί με την σχεδίαση για την εξυγιανσιμότητα του SRB, του Συμβουλίου Εξυγίανσης, θα πρέπει να βοηθήσει να φέρουν τις τράπεζες σε μια δυνατότητα να αντιμετωπίσουν όλα τα αδύνατα σημεία τους όπου υπάρχουν δυσκολίες εξυγίανσης και όπου δεν ξέρετε πού θα μπορέσουν να βρουν το κεφάλαιο για να αντιμετωπίσουν τις εκθέσεις του. Καλή συνεργασία λοιπόν μεταξύ των υποπτικών αρχών και των αρχών εξυγίανση για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά από κοινού. Σα ευχαριστώ. Ο κ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξέρω πώς, αντιμετωπίζετε την τωρινή κατάσταση στα ευρωπαϊκά πιστοτικά ιδρύματα. Δηλαδή, τι κίνητρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες, κατά την άποψή σας, παίρνουν ακόμα και τώρα, αναλαμβάνουν κινδύνους ε, ε υπερβολικούς, ακόμα και τώρα γιατί πιστεύουν θα τους διασώσουν τα κράτη, ο δημόσιος τομέας και θα λέγατε ότι είναι υποκεφαλαιόμπε, υποκεφαλαιοποιημένες, γιατί έδειξαν κάποιες δυσκολίες στα, οι αντοχής. Εσείς λέτε ότι φταίει ότι είναι η κρίση που το έχει οδηγήσει αυτό, αλλά μήπως είναι και αποτέλεσμα της εντύπωσης ότι θα τους σώσει ο δημόσιος τομέας. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό τουλάχιστον. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. με το γεγονός ότι πράγματι σε κάποιο βαθμό η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση έχει αλλάξει τις συνθήκες του παιχνιδιού. Το βλέπετε και αυτό από, αν κοιτάξετε, εξωτερικές αξιολογήσεις των τραπεζών αυτό. Οι εταιρείε πιστοληπτικής αξιολόγησης έχουν βγάλει το κομμάτι της λεγόμενης κρατικής κυδαιμονίας σε ό,τι αφορά το, την αξιολόγηση του κινδύνου. Στο βαθμό αυτό <clears throat> θα σας έλεγα ότι αν δούμε τώρα την κατάσταση όπως έχει και φυσικά υπάρχει το λεγόμενο home bias, υπάρχει το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη ε, ναι, ένα είδος μεροληψίας προς, τους, ε, προς τους εγχώριες δραστηριότητες. Σίγουρα δεν βρίσκονται όλες οι τράπεζες εκεί που θα πρέπει να βρίσκονται υπό την έποψη της ε, εξυγιανσιμότητος και ίσως χρειαστεί, όπως είπατε, και κάποιος χρόνος για να φτάσουν εκεί. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σαντ θέλει και πάλι το λόγο. Κυρία Κένικ είσαστε ικανοποιημένοι με την αρχιτεκτονική της Τραπεζικής Ένωσης και κυρίως με τις εξησίες και τις αρμοδιότητες του μηχανισμού εξυγίανσης. Μήπως θεωρείτε ότι είναι απόρρια πολιτικών συμβιβασμών, παραδείγματος χάρη. Οι αρμοδιότητες για την παρέμβασή σας είναι πολύ περιορισμένες στη Γερμανία αν τη συγκρίνουμε με τις δυνατότητες σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία. Μήπως θα ήταν καλύτερο να υπάρχει συγκρισιμότητα εξουσιών και αρμοδιοτήτων. Και πόσο είσαστε πεπισμένοι ότι τα πολιτικά κριτήρια δεν θα επηρεάσουν αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται από το Συμβούλιο Εξήγησης. Αν φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, πιστεύετε ότι θα υπάρξει ίδια αντιμετώπιση για τις μικρές τράπεζες της Μάλτας της Κύπρου και άλλοι για τις μεγάλες τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας. Και πιστεύετε ότι θα υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ του, ε, Ταμείου Εξυγε... του Συμβουλίου Εξυγίανσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πώς μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια συνεργασία για τις αρμοδιότητες παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε δει όλοι στα μέσα ενημέρωσης ε, παρουσίαση των μηχανισμών αυτών. Εγώ είμαι πραγματίστρια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα, μπορεί κάποτε να υπάρξει μια αναθεώρησή τους όταν οι πολιτικοί ηγέτες αποφασίσουν ότι μπορούν να βελτιωθούν. Αλλά για να είμαι δίκαια σε σχέση με αυτό που είπατε, αυτό ακριβώς τονίζει τη σημασία του να Προσπαθούμε να είμαστε προδραστικοί, να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ε, εξυγιανσιμότητα και να μην περιμένουμε το Σαββατοκύριακο που θα γίνουν όλα, όπως λέμε. Για την πολιτική πίεση, ότι μπορεί να έχει διαφορετικό αντίκτυπο για τις μικρές ή τις μεγάλες χώρες ή τις μικρές τράπεζες έναντι των μεγάλων όλοι είμαστε δεσμευμένοι στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και στην ισότητα ανταγωνισμού, για μένα σημαίνει αναλογικότητα και στη σχεδίαση της εξυγίατσης. Δεν χρειαζόστε τα ίδια σχέδια για μια μικρή και λιγότερο πολύπλοκη τράπεζα, όπως αυτά που θα χρειαστείτε για μια μεγάλη τράπεζα, αλλά σαφώς το σύστημα θα πρέπει να ισχύει για όλους, και ακόμα και ιδίω αν πρέπει να υπάρξει εξυγίανση μιας τράπεζας. Είναι δύσκολο εγώ βέβαια να κάνω κάτι το οποίο δεν θα είναι λογικό. Και το τελευταίο σας ερώτημα. Αναφερθήκατε στο ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό για το μηχανισμό εξυγίανσης να είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, μια ευρωπαϊκή φωνή σε αυτή τη συζήτηση η οποία μπορεί να είναι τεχνικού χαρακτήρα για να επιληθούν τα προβλήματα της εξυγίανσης, ιδίως τα διαμεθοριακά εμπόδια εξυγίανσης όταν πρόκειται για επιχειρήματα ότι αυτό δεν δουλεύει καλά ή εκείνο δεν δουλεύει καλά και κάποιοι έχουν κάποιες προτάσεις, λύσεις. Εγώ συνήθως ακούω τις καλές ιδέες και ελπίζω ότι και όλο το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα έχει μια σαφή άποψη για το πώς θα προχωρήσουμε και να δούμε τι θα πετύχουμε έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι κάνει άμα βρεθεί σε τέτοιες δύσκολες περιστάσεις. Ευχαριστώ. Ο Μπράιν Χέις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Τρεις σύντομες ερωτήσεις Πρόεδρε. Θα μπορούσατε να μας κάνετε μια σύντομη περιγραφή του επίπεδου συνεργασίας ανάμεσα στο SSM και το δικό σας όργανο Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να συνδεθείτε, να συνεργαστείτε γιατί υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα ε, το οποίο έχει δημιουργήσει μέσω των stress tests ε, και ίσως να κάνω λάθος αλλά είχα πει ότι οι χώρες ε, της εκτός Ευρωζώνης θα συνδεθούν ε, με το SSM γιατί νομίζω ότι θα γίνει το διεθνές επίπεδο αν θέλετε και σε επίπεδο και ύψους κεφαλαίων και γενικότερα για τα πιστοτικά ιδρύματα. Uh, το Ταμείο Εξυγίανσης λοιπόν, η πρόσβαση σε πιστώσεις θα γίνει από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα χρήματα θα δίδονται ε, επί τούτου κάθε φορά όποτε χρειάζεται. Και τέλος γνωρίζετε το επιχείρημα για τη μετάβαση που έχουν ορισμένοι προτείνει ότι ανάμεσα στο σήμερα δηλαδή και στην πλήρη ταχύτητα λειτουργίας θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι συνεισφορές των διαφόρων χωρών. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό σχετικά με την συνεργασία ανάμεσα στο SSM και στο δικό μας όργανο είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ στενή συνεργασία. Ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας είναι υπεύθυνο για την εποπτεία αλλά είναι ταυτόχρονα υπεύθυνο είναι το πρώτο όργανο αν θέλετε ε, στο οποίο θα απευθυνθεί μια τράπεζα όταν κινδυνεύει να αποτύχει ή όταν έχει ήδη αποτύχει. Ελπίζω λοιπόν γνωρίζοντας τον Τανιέλ Λουί και γνωρίζοντας πως ε, το ταμείο αυτό θα, η αρχή αυτή θα λειτουργήσει ε, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να παρεμβαίνουν ακριβώς επειδή κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ε, απαιτείται μια πολύ στενή συνεργασία λοιπόν και για τα θέματα της ανάκτησης ε, των ε, πιστοτικών δραστηριοτήτων και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός εδώ, ιδιαίτερα όταν ερχόμαστε σε επαφή με τις τράπεζες οι οποίες θέλουν καθοδήγηση σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Εγώ λοιπόν περιμένω να υπάρξει μια στενή και πολύ καλή συνεργασία. Ε, σχετικά τώρα με το Ταμείο Εξυγίανσης. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε νωρίτερα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε την ικανότητα για το συγκεκριμένο ταμείο να δανείζεται ή να έχει εν πάση περιπτώσει μια δυνητική δυνατότητα δανεισμού. Αυτό ε, θα ε, του επιτρέψει ε, να κρίνει αν θα αναζητήσει χρήματα από το εθνικό επίπεδο ή από το κοινοτικό επίπεδο ή από την ιδιωτική αγορά ή από ονδήποτε ο οποίος θέλει να πάρει μέρος στην διαδικασία αυτή δανειοδότησης. Όπως και το προβλέπει ο κανονισμός στα πλαίσια της λειτουργίας των λογωμένων backstops. Η τελευταία σας ερώτηση δεν την συγκράτησα, μπορείτε να την επαναλάβετε. Νομίζω ότι από ό,τι το βλέπω εγώ, το 2015 θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το Ταμείο μας όπως ε, και το 2014 ήταν αυτό που υπολογίσαμε για το SSM. Θα πρέπει όμως τα χρήματα αυτά να τα δαπανίσουμε με σωστό τρόπο, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Από τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα και σε εθνικό επίπεδο και σε συνεργασία με άλλες εθνικές αρχές, ότι μιας και τώρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, θα πρέπει να αποφασίσουμε πρώτα την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και αν και μιας και έχουμε αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα για την ενιαία εποπτεία, έχουμε και το θέμα της ανάκτησης των τραπεζών, το οποίο έχουμε σχετικά ορίσει. Σε συνεργασία λοιπόν να τα συζητήσουμε αυτά με τις εθνικές αρχές και θα πρέπει επίσης ε, να γνωρίζουν και οι τράπεζες ε, τι μπορεί να τις ε, περιμένει και να γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθηθούν. Εγώ δεν, δεν έχετε κανένα πρόβλημα σε σχέση με την έννοια της μεταβατικότητας. Εγώ αναφέρομαι στην μετάβαση, αν θέλετε, από από το εθνικό επίπεδο σε κοινοτικό επίπεδο. Για τη μεταβατικότητα των πληρωμών απαιτούνται περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ δεν είμαι κατά αυτής της μεθόδου. Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε το θέμα και από απόψεως ρευστότητας και από απόψεως κεφαλαίου. Δεν θέλει κανείς να βρεθεί σε με τέτοια θέση όπου αν χρειάζεται τα χρήματα κάποιος να πει όχι είναι πολλά γιατί δεν τα είχαμε προγραμματίσει. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορεί να είναι κανένας προκυκλικός, από την άλλη τίθεται και το κατανοώ το θέμα της ρευστότητα. Νίνα Τζίλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δόκτωρα Κέρνιγκ, ε, σημαντικές μεταρρυθμίσεις έγιναν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ωστόσο παραμένει το πρόβλημα των πολύ μεγάλων ε, τραπεζών, too big to fail. Η αυτές που είναι πολύ πολύπλοκες για να γίνει εξηγένσή τους. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι κάποιες τράπεζες συνεχίζουν εμέσως να επιδοτούνται με χρήματα των φορολογουμένων. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς το πρόβλημα αυτών των too big to fail τραπεζών, πώς θα το αντιμετωπίζετε και για τις τραπεζικές διαθωτικές μεταρρυθμίσεις και το διαχωρισμό τραπεζών, ποια είναι η άποψή σας. Πρώτη ερώτηση αυτή και δεύτερη, σε περίπτωση Σοβαρή συστημική κρίση. Το πρόβλημα της εξυγίανση ε, μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομήλων θα είναι ιδιαίτερως δυσχερέ, ιδίω από τη στιγμή που στην Ευρώπη δεν υπάρχει συμφωνία για δεσμευτικό μηχανισμό διαιτησία για την ε, εξυγίανση τραπεζών, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Πώς θα προβείτε λοιπόν στην εξυγίανση μιας μεγάλη και συστημική συστημικής τράπεζας, η οποία δραστηριοποιείται υπό διαφορετικά εποπτικά καθεστώτα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και ε, υπό το πρίσμα του προβλήματος που έχουμε για την ε, επίλυση του προβλήματος ε, των τραπεζών όπως η Φόρτις και άλλων. Απάντηση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι οι πιο μεγάλες τράπεζες και δεν μιλάω μόνο για την Ευρωζώνη, αλλά για όλο τον κόσμο, εάν πρέπει να εξηγενθεί μία από αυτές τις τράπεζες τέτοιου μεγέθους, JP Morgan, Barclays, ε, Deutsche Bank κτλ, πάντοτε και κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργείται τα πια αναταραχή και κάποιο κενό. Βέβαια δεν υπάρχει άλλη λύση, αν δεν υπάρχει μάλλον τέτοια λύση, Ιδίως αν δεν έχει τράπεζα ένα στέρεο σχέδιο καταρχάς ανάκαμψης ε, και κατά δεύτερον εξυγίανσης. Άρα τότε δεν θα υπάρχει άλλη λύση. Και υπάρχουν και τα διαρθρωτικά, τα δομικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η έκφραση too big to fail ε, πάντα εστιάζουμε πολύ στο μέγεθος, αλλά εγώ θα έλεγα πρέπει να τονίσουμε και το too complex ή ε, το, το, της πολυπλοκότητας της οργάνωσης δηλαδή. Γιατί εκεί έκειται το θέμα. Η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και ο, καθο... ο για το μηχανισμό εξυγίανσης μας δίνουν εργαλεία. Είπατε όμως και κάτι σημαντικό που δεν έχουμε βρει γι' αυτό ακόμη λύση. Δηλαδή, όλες αυτές οι τράπεζες που αναφέρατε εργάζονται σε παγκόσμια κλίμακα, το είπα και εγώ πριν. Δεν έχουμε όμως ένα παγκόσμιο ρυθμιστή. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσουμε το ίδιο μονοπάτι που έγινε και σε εθνικό επίπεδο και από άλλους φορείς. Δηλαδή, για θέσεις τράπεζες έχουμε τους ομίλους διαχείρισης κρίσεων. Οι βασικές δικαιοδοσίες ε, προορισμού και υποδοχής ε, εξεργάζονται το κοινό σχέδιο εξυγίανσης και πρέπει να συμφωνήσουν και για τη χρηματοδότηση των διαφορετικών κομματιών του ομίλου. Δεν μπορεί να ισχύει σε μικρότερη και σε μεγαλύτερη κλίμακα, διότι αν πραγματικά φτάσουμε σε μια κρίση, εγώ πιστεύω πιο πολύ στην εμπιστοσύνη μεταξύ των ρυθμιστών. Για τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες, ε, το SRB Δηλαδή θα πρέπει να μπορεί να ε, λύσει το ζήτημα προ ε, προς όφελος των ομίλων. Αλλιώς καταστρέφεται η στρατηγική της εξυγίανσης. Ευχαριστώ. Είσαστε έτοιμοι λοιπόν να μπείτε σε, αυτό το, σε την ομάδα εργασίας για τη διαχείριση των κρίσεων. οι, ομάδες, οι επιτροπές εξυγένσης θα πρέπει να δημιουργηθούν ούτως ή άλλως, αλλά για τις μεγαλύτερες τράπεζες πρέπει να είναι οι ομάδες διαχείρισης κρίσης, γιατί πρέπει να συμμετάσχουν και οι άλλοι φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε Πολιτείε είπαν ότι κάνανε κάποια ε, αν θέλετε, εξομοίωση για τέτοιες περιπτώσεις, ένα παιχνίδι πολέμου, αλλά προς όφελος της ειρήνης. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ξέρει ο καθένας πώς θα αντιδράσουν οι άλλες πλευρές και θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη εμπιστοσύνη μεταξύ των ρυθμιστών ή καλύτερα μεταξύ των αρχών εξυγίανσης. Ο Μπέρντ Λάγκε, Βέρνερ Λάγκε, συγγνώμη. Κυρία Κιόνιχ, ε, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση της ικανότητάς σας και αυτά είναι θέματα τα οποία βέβαια είναι υπό επεξεργασία και γι' αυτό παραμένουν κάποια θέματα ανοιχτά. Εσείς ως πρόεδρος της Μπάφιν είσαστε μέρος της Επιτροπής της, Βασιλεία, της Βασιλείας η οποία έχει επικρίνει την προηγούμενη εβδομάδα κάποια τμήματα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας εξαιρέσεις για την ε, αντιμετώπιση των ε, παραγόγων. Αυτό αντιμετωπίστηκε αρνητικά. Επίσης οι αξιολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική ικανότητα έχουν ε, τύχει επικρίσεως, αλλά και η αντιμετώπιση του κρατικού χρέους επίσης. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς κρίνετε εσείς εν γέννη τις ρυθμίσεις, τις αποφάσεις που έχουμε πάρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Είναι υπερβολική η ρύθμιση όπως λένε οι ενδιαφερόμενοι είναι κάτι το οποίο αποκλίνει από τις ρυθμίσεις των ε, Ηνωμένων Είναι κάτι το οποίο συνάδει με τις ρυθμίσεις της Βασιλείας ή όχι. Σας ευχαριστώ για την φιλοφροσύνη σας. Μπορώ να είμαι σύντομη. Αυτό μπορώ να σας απαντήσω ότι ο αρμόδιος διευθυντής για την εποπτεία των τραπεζών θα είναι μέλος της Επιτροπής της Βασιλείας. Εγώ δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής πια. Αλλά φυσικά η Επιτροπή της Βασιλείας έκανε επικρίσεις αλλά είπε ότι αυτά είναι μικρά πράγματα. Οι επικρίσεις λοιπόν που έχουν δημοσιευθεί ίσως είναι υπερβολικές. Υπάρχει το θέμα του κρατικού χρέους και της αντιμετώπισης του στους ισολογισμούς των τραπεζών, αλλά εν γέννη κάθε χώρα έχουν, δίδουν μηδενικό ε, ρίσκο για το δικό τους εθνικό κρέος. Αλλά δεν θέλω τώρα να μπω σε τεχνική συζήτηση. Εγώ αποδέχομαι ότι δεν υπάρχουν χρέη τα οποία έχουν μηδενικό κίνδυνο. Και φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του κρατικού χρέους κάποια στιγμή τα άλλα σημεία τα οποία είπε η Επιτροπή της Βασιλείας. Ναι, υπάρχουν διαφορές με τις ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν και αποχρόντες λόγοι για αυτή τη διαφορά. Το βασικό σας θέμα είναι πώς βλέπω εγώ εν γέννη αυτό το ζήτημα. Εμείς ερχόμαστε από μια φάση απορρίθμισης μετά από την ε, χρηματοπιστική κρίση. Περνάμε σε άνα επαναρρύθμιση των θεμάτων των τραπεζών και νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει τους βασικούς δομικούς λίθους για αυτήν την επαναρρύθμιση στον πιστοτικό τομέα. Στους τομείς των μη τραπεζικών πιστοτικών ιδρυμάτων υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Τα θέματα των ε, χρηματιστηρίων και των τόπων συναλλαγής και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία εξυγένσης. Αλλά πιστικά αρχίζουμε να περνάμε στη, βάση, στη φάση της ε, εφαρμογής και της εποπτείας της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Και γι' αυτό νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει να πει η Επιτροπή της Βασιλείας είναι πρέπει όλοι αυτοί οι κανόνες ταυτόχρονα να εφαρμοστούν σωστά. Ευχαριστώ. Δύο συνάδελφοι ζητήσανε να λάβουν το λόγο στη διαδικασία κασία και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Κλείνω τον κατάλογο αγορητών. Ο Μπεντ Λούκε και ο Φάμπιο Δεμάση θα λάβουν το λόγο κυρία Κιόνικ. Επανέρχομαι σε ένα προηγούμενο ερώτημα. Ξέρω ότι ο κάθε επενδυτή είναι τελικά και αυτός φορολογούμενος. Αλλά υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι επενδύσεων, διάφορα επενδυτικά σχήματα. Υπάρχουν τα ταμεία ασφαλίσεως, ε, τα ασφαλιστικά ταμεία, συγγνώμη, τα συνταξιοδοτικά ταμεία ε, αυτά τα οποία εξασφαλίζουν την ε, ε, σύνταξη παραγωγικά των πολιτών. Υπάρχει εδώ πέρα, είναι, μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα που έχουν αυτοί οι τομείς. Εγώ δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένες τράπεζες, αλλά συνολικά πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και πώς θα πρέπει να κινητοποιηθούν σε μια περίπτωση bail-in. Αυτό είναι κάτι το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να πει κάτι σε σχέση με όλα αυτά και γι' αυτό θέλουμε να μας πληροφορείτε σχετικά. Ίσως έχω παρακάμψει το σημείο αυτό λέγοντας. Υπάρχει πράγματι μια σκέψη η οποία θα πρέπει να δοθεί για το ερώτημα του πώς τα, κεφάλαια αυτά τα οποία είναι τα πιο εκτεθειμένα να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση bail είναι. Και εδώ τίθεται το θέμα του αν κατέχει μια τράπεζα το κεφάλαιο αυτό το οποίο έχει σε στόχο την απορρόφηση κινδύνου μιας άλλης τράπεζας. Και τι γίνεται όταν η τράπεζα αυτή μπαίνει και αυτή σε δυσκολίες. Νομίζω ότι αυτή τη σκέψη όμως θα πρέπει να την ε, λάβουμε μαζί με μια πρέζα αλάτι όπως λέμε και για τους άλλους επενδυτές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επομένως την κατάσταση που μπορεί να προκύψει για τους άλλους επενδυτές και αυτό είναι ένα θέμα ρύθμισης το οποίο προφανώς θα πρέπει να συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μένα δεν είναι επομένως η λύση να εξαιρέσουμε συγκεκριμένους επενδυτές από τη διαδικασία του bail αλλά απλώς να καθορίσουμε το μέγιστο ποσό στο οποίο μπορούν να κληθούν να συμβάλλουν αυτοί οι ευαίσθητοι επενδυτέ στη διαδικασία του Μπέιλιν. Ο Φάμπιο Ντεμάζη. Και το δικό μου ερώτημα. Α, στα αγγλικά. Στα αγγλικά για να ακούσετε διαφορετικές γλώσσες και να μην βαριώσετε, να μην νομίζετε ότι είναι καθαρά γερμανική υπόθεση. Ή και ιταλικά μπορώ να το πω. Είπατε ότι υπάρχουν ε, στον μη στο μη τραπεζικό τομέα ορισμένα κενά. Ο μη πιστοτικός τομέας, ο σκιώδης πιστοτικός τομέας, όλα αυτά διαφεύγουν αυτή τη στιγμή κοινοτικού ελέγχου. Και αναφερθήκατε λίγο σε αυτά. Αλλά σχετικά με τα phasing out, Ποια είναι η άποψή σας γύρω από αυτό και τι πιστεύετε Same prudential regulations as banks. Um, Νομίζω ότι τα σύναψη λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι τράπεζες. Δεν θα πρέπει να κάνουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτή είναι η θέση την οποία έχουμε γενικότερα. Νομίζω ότι η θέση ε, για τα ΣΥΝΑΒ και τις αγορές των νομισμάτων ε, δεν είναι να αποκτήσουν τραπεζική άδεια, αλλά να υπόκεινται στους, δύο, στους ίδιους μηχανισμούς με τον τραπεζικό τομέα. Και εδώ σας μεταφέρω τη δική μου άποψη είναι δύσκολο να κατανοήσω την λογική πίσω από ένα ταμείο σύναφ αν είναι έτσι και αλλιώς ένα κομμάτι ένα συστατικό ενός ταμείου που έχει κειμενόμενη έτσι και, αλλιώς, έτσι και αλλιώς αξία. και θα έλεγα ότι τα ταμεία ακριβώς είναι κεντρική αντιβαλόμενη δηλαδή από τη μία έχουν συναλλαγές σε μια οργανωμένη και αναγνωρισμένη πλατφόρμα από την άλλη όμως τίθεται ένα θέμα συστημικό εδώ. Είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις και αν κάποια από αυτές απτοκεύσει, αποτύχει, το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο πιθανής ανάκτησης ή μάλλον η ανάκτηση είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει αλλά πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εξυγένσης. Thank you. Mr. Langen for very quick follow-up. Λοιπόν, ο κύριος Λάγκεν, συμπληρωματική ερώτηση. Για τους ε, CCPs, για τα κεντρικά αποθετήρια, μάλλον για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, έχουμε για τα παράγωγα καθορίσει ορισμένε. Ε, εξαιρέσεις για τα παράγωγα τα οποία έχουν συγκεκριμένο στόχο εξασφάλισης και έχει αναφερθεί ότι για τα τα ταμεία θα υπάρξει μία εξαίρεση για τρία χρόνια. Αλλά σε αυτά τα τρία χρόνια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση. Και η Κομισιόν θέλει να τα εξαιρέσει από προς το παρόν από τη συζήτηση για τα παράγωγα. Θα ήθελα να έχω την άποψή σας και την κρίση σας για τα θέματα αυτά. Εγώ δεν ξέρω πολλά για αυτά τα θέματα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν μπορώ να σας δώσω μια τεκμηριωμένη απάντηση, αλλά είμαι έτοιμη να μάθω περί τίνος πρόκειται και να επανέλθω ενώπιον σας. Σας ευχαριστώ, Δόκτωρ Κούνιχε για την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Όπως ξέρετε θα σταματήσουμε. Θα περατώσουμε μάλλον την ακρόαση των άλλων μελών. Αύριο το πρωί ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 15 Δεκεμβρίου και στις 16 στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ και τελειώνει η συνεδρίαση και τα σκουλαρίκια.